Okay, colleagues, I think we're Να ξεκινήσουμε, συνάδελφοι. Έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες, ε, πολλές, ε, ε, πολλές συμβιβαστικές, επομένως. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα όμως να καλεσορίσω δύο ομάδες καθηγητών εξ ονόματος του καθηγητού Κανοντεύσκη. Θα ήθελα να καλωσορίσω μία ομάδα που έχει προσκαλέσει. Είστε εδώ. Από τον κύριο Κασνοντεύσκη καλεσμένοι να σας καλωσορίσω και επίσης έχουμε ε, και μία ομάδα από το δίκτυο των πόσκο που δουλεύει με παιδιά για την καταπολέμηση της φτώχειας, με νέους ανθρώπους. Ε, η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ είναι πολύ σχετική με τη δουλειά που κάνετε και εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε στην ομάδα μας. Πριν αρχίσουμε την ψηφοφορία, να κάνουμε μια δοκιμαστική <clears throat> ψηφοφορία για να δούμε αν είμαστε όλοι εδώ. Έχουμε 20 ψηφίζοντες. Λειτουργούν όλα, πάρα πολύ ωραία, όλες οι κάρτες ε, λειτουργούν, είμαστε 21. Πολύ ωραία η δοκιμή λοιπόν πέτυχε, ξεκινάμε με τις πολιτικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Λατινική Αμερική. Ενρίκε είναι ο εισηγητή. Ενρίκε, θέλεις να πεις κάτι πριν ξεκινήσουμε. Όχι, θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω τις πολιτικές ομάδες για την καλή συνεργασία σε σχέση με τούτη τη γνωμοδότηση. Νομίζω ότι ε, ε, μεταξύ Στρασβούργου, Τυρκουάζ εβδομάδων, ε, δυσκολιών διαφόρων, καταφέραμε παρόλα αυτά να βρούμε συμβιβαστικές τροπολογίες και εγώ προσπάθησα να υποβάλω συμβιβαστική λύση σχεδόν για κάθε μία από τις παραγράφους του σχεδίου γνωμοδότησης. Ευχαριστώ όλους για αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινούμε λοιπόν με τη συμβιβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός ε, Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 ε, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα της τροπολογίας 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται παρόλα αυτά καλύτερα να ε, κάνουμε μια επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Από τις τροπολογίες 29. Πέρας. Και εγκρίνεται όντως. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω πως εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να κάνουμε μια επαλήθευση για την τροπολογία 43, άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές Καλύτερα να το επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα αυτό. Ε, τροπολογία 47. Πέρας και εγκρίνεται. Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 κατά τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Όχι, συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος 66. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του συνόλου. Άρχεται η ψηφοφορία. Διονομαστικής κλήσεως η Πέρας και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία 17 ψήφοι υπέρ, 5 ε, αποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την προσπάθεια που κάνατε να βρείτε συμβιβαστικέ λύσεις. Πολύ ωραία. Okay, we move on now to the... Περνάμε τώρα στην επόμενη γνωμοδότηση σχετικά με τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιωσιμότητα. Ε, είναι το δίδυμο κείμενο κατά κάποιο τρόπο για, ε, σε σχέση με το άλλο κείμενο για, την, ε, για τους στόχους βιωσιμότητας. Θέλετε κυρία Σλάιν να πείτε κάτι πριν ξεκινήσουμε. Όχι να ευχαριστήσω μόνο όλους τους σκιώδεις ηγητές για την πολύ καλή συνεργασία και δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ έχουμε, λέει η Πρόεδρος, πολλές συμβιβαστικές. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά 8, ε, συγγνώμη, κατά εγκρίνεται, συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές ε, καλύτερα να επαληθεύσουμε. Τροπολογία 36, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 37, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 38, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 48, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές ε, θα ελέγξουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 49 πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 77. Πέρας της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, είμαι σίγουρη ότι έχει εγκριθεί, αλλά παρόλα αυτά καλύτερα να το ε, ελέγξουμε πέρα της ψηφοφορίας. Ναι, έχει εγκριθεί. Τροπολογία 82. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, ε, συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω πως έχει απορριφθεί, αλλά καλύτερα να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε και απεριφθεί. Ε, ψηφο, ψηφοφορίες από τον αιτιολογικών σκέψεων, συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροποποιημένη γνωμοδότηση με ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια, Έλλη Σλάιν. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη γνωμοδότηση αυτή. Τώρα ψηφίζουμε για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως για τη διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα στις τρίτες χώρες. Σκληρή δουλειά από μεριά του συναδέλφου μας, του κύριου Στέλιου Κούλογλου, που είναι εδώ κοντά μου, δίπλα. Θέλετε να πείτε τίποτα κύριε Κούλογλου, όχι. Άλλωστε τα είπαμε μόλις χθες. Ήταν μια θετικότητα τη συζήτηση χθες. Αρχίζουμε λοιπόν με τη συμβαστική 1. Παρακαλώ ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε νομίζω ότι εγκρίνεται Α, όχι όχι σαφώς, σαφώς, σαφώς εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα της 18 υπέρ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 κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα της 28 α όχι αυτό εκπίπτει ακολουθεί μια χωριστή ψηφοφορία επί του αρχικού ψηφίζουμε ξεχωριστά την αρχική παράγραφο 6 ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουν αποσυρθεί οι δύο τροπολογίες κυρία Στόια. Ψηφίζουμε λοιπόν ονομαστικά το σύνολο της ε, γνωμοδότηση. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται και μάλιστα ομόφωνα. Συγχαρητήρια, αγαπητέ Στέλιο. Και σας ευχαριστώ όλες και όλους. Okay, the next, the next... Ευχαριστώ. Λοιπόν, η επόμενη ψηφοφορία είναι επί του σχεδίου γνωμοδοτήσεως για τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ε, Ένωσης της Παγκόσμιας Αλυσίδας Αξίας. Ιγνάσιο, επιθυμώ να ευχαριστήσω τους και όλους τους και εισηγήτριες για την συνεργασία. Μάλιστα, πρόκειται για γνωμοδότηση για, η οποία θα απευθυνθεί στην, στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου.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 ομόφωνα δεκτή. Συγχαρητήρια αγαπητέ Ιγνάσιε. Και μάλιστα με μεγάλη συνέντευξη. Πολύ ωραίο αυτό, διότι όλοι συμφώνησαν με όλα σχεδόν. Και τώρα ερχόμαστε στην τελευταία ψηφοφορία. Έχει γίνει πολλή δουλειά στις ε, συμβαστικές. Πρόκειται για σχέδιο γνωμοδοτήσεως που θα απευθυνθεί στην Επιτροπή ΙΝΤΕ για τον πολιτικό διάλογο και την συμφωνία συνεργασίας με την Κούβα με εισηγητή τον κύριο Φρανκ Έγγελ τον οποίο καλό αν θέλει να λάβει το λόγο. Μια μισή φράση μόνο κυρία Πρόεδρε. Εν ώψη του γεωγραφικού προορισμού του κειμένου αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξαν κάποιες ιδεολογικές διαφορές ανάμεσα στις τοποθετήσεις των μεν και των δε και βέβαια θα γίνει έχουμε να ψηφίσουμε αρκετά πράγματα, παρόλο που το κείμενο συνολικά είναι μόνο μια μισή σελίδα. Είναι σημαντικό πάντως ε, να πούμε ναι στη συμφωνία αυτή, γιατί για πρώτη φορά γίνεται τέτοια ε, σημαντική συμφωνία με την ε, χώρα αυτή, την Κούβα δηλαδή. Η πρόεδρος. Ψηφίζουμε πρώτα το ψήφισμα και μετά θα ψηφίσουμε για τη συνένεση. Αρχίζουμε λοιπόν με το ψήφισμα. Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Τροπολογία 3. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Τροπολογία 7. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την τροπολογία 20. Νομίζω όμως ότι απορρίπτεται. Πέρας. Α, εγκρίνεται. Συγγνώμη, μου φάνηκε ότι οι ορισμένοι απήχαν. Τώρα 21 χωρίζεται σε δύο τμήματα. Okay, so very quick. Okay, we'll do it for longer. And yeah. Okay, we're okay, we'll, we'll do it slowly. We'll do it slowly. It will... Okay, θα κινηθούμε ε, αργά. Τροπολογία 21, η οποία χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα τώρα, υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση στο σύνολό της με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Πέρας. Και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. έχει καλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ βεβαίω και τον κύριο Έγγελ. Τελειώσαμε. Α, όχι, όχι, όχι, συγγνώμη, έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό ακόμη. Βεβαίω, το πιο σημαντικό κατά κάποιο τρόπο. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα. Ψηφίζουμε περί της συνένεσης χωρίς τροπολογίας. Ψήφι Α, με συγχωρείτε, πρέπει να είναι ηλεκτρονική η ψηφοφορία αυτή. Δηλαδή ονομαστική. Ε, αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή. λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ Έγγελ για τις δύο εκθέσεις. Και μάλιστα τώρα τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας. Okay, colleagues, we, we actually finished votes very early. We have... Συνάδελφοι, τελειώσαμε γρήγορα τις ε, ψηφοφορίες, γιατί θέλαμε να αφήσουμε και ένα περιθώριο χρονικό ε, για τις ε, τροπολογίες που θα καταπίπτουν. Αυτό σημαίνει όμως ότι οι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν καταφτάσει ακόμα. Ένα μικρό διάλειμμα λοιπόν 10-15 λεπτών μπορείτε να πάτε να πάρετε καφέ.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

Συνάδελφοι, συγγνώμη για την ε, καθυστέρηση. Περιμένουμε τους ε, καλεσμένους μας, γιατί ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες ε, νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Καθίστε λοιπόν, παρακαλώ. Um, so it's item 17. Λοιπόν, σημείο 17 η αξιολόγηση των μηχανισμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το συνδυασμό δανείων με επιχορηγήσει. θα έχουμε παρουσίαση από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την έκθεση με θέμα τη διευκολύνσης τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για το συνδυασμό δανείων και επιχορηγήσεων ω μηχανισμό για την παροχή βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντική αυτή η διαδικασία γιατί βρισκόμαστε εν μέσω τριμερών διαλόγων ακριβώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξη που θα συμπληρώσει οι ε, ε, υποδομές ε, για το συνδυασμό δανεισμού και επιχορηγήσεων. Ο συνδυασμός είναι ένας τρόπος παροχής επιχορηγήσεων ως μηχανισμό μόχλευσης δανεισμού για μεγάλες επενδύσεις αρκεί να υπάρχει εγγύηση επιστροφής και απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαμορφώσει 8 ε, τέτοιε ε, διευκολύνσεις ε, που καλύπτουν το σύνολο της εξωτερικής βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντική χρηματοδότηση. 2,3 δι ευρώ έχουν κατανεμηθεί εκεί από το 2014 για μια επταετή περίοδο. Το 2014 υπήρξε μια έκθεση που έλεγε ότι είναι αποτελεσματικός αυτός ο μηχανισμός, αλλά υπήρχαν και κάποιες κριτικές για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων ε, και τις διαδικασίες απονομής των επιχορηγήσεων, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για την ε, ε, αξία των επιχορηγήσεων. Υπήρξε μια εξωτερική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το τύπο βοήθειας και περί αυτού θα γίνει η σημερινή παρουσίαση. Είχαμε και την συμβουλευτική, ε, την, υπηρεσία, την ε, εταιρεία παροχής ε, υπηρεσιών ADE. Σήμερα θα ακούσουμε από τον κύριο Έντριαν Κωνσταντάτσε, από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, από την Μονάδα αξιολόγηση, και θα μας δώσει τα βασικά πορίσματα της έκθεσης, τα οποία έχουν παρουσιαστεί και στα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο ενός ειδικού σεμιναρίου. Ο κύριος Καϊπακλής επίσης είναι εδώ, επικεφαλής ε, της μονάδας και μπορεί ενδεχομένως να προσθέσει δύο πράγματα. Παρακαλώ, κύριε Κωνσταντάτση. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία αυτή να σας παρουσιάσουμε σήμερα ε, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που εκπονήσαμε όπως ανέφερε και η Πρόεδρος, αυτή η αξιολόγηση έχει γίνει από μια ομάδα ανεξάρτητων αξιολογητών και η μονάδα αξιολόγηση την οποία εκπροσωπώ έχει συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία. Το αντικείμενό μας ήταν το blending, ο συνδυασμός λοιπόν αυτός, ε, που είναι μια μορφή χρηματοδότησης ε, συνδυάζοντας ε, δάνεια με επιχορηγήσεις. Και αυτό δεν γίνεται μόνο για να ε, συνδυάσουμε διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης, αλλά επειδή υπάρχει μια σειρά ωφελών που θεωρούμε ότι έτσι προκύπτουν. Αυτά τα ωφέλη περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ε, την αύξηση της δυνατότητας βιωσιμότητας αυτών των ε, έργων και έτσι την προσέλκυση επενδύσεων, βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας ε, και της βιωσιμότητας των έργων που επιδοτούνται, την αύξηση της προβολής και της διαφάνειας ό,τι αφορά τις δαπάνες, το κόστος αυτών των έργων, αλλά και ένας πιθανός αντίκτυπος στις πολιτικές που διαμορφώνονται μετά τα έργα. Η αξιολόγηση καλύπτει 7 από τις 8 ε, διευκολύνσεις ε, που μέχρι το 2014 ε, είχαν χρηματοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και η περίοδος αξιολόγησης είναι 2007 έως 2014. Γενικά η αξιολόγηση είναι θετική σε ό,τι αφορά το blending και καταδεικνύεται ξεκάθαρα η σημασία του μηχανισμού, παρότι υπάρχουν αδυναμίες και προκλήσεις, γενικά βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά. Η αξιολόγηση δομήθηκε γύρω από τρεις βασικούς ε, πυλώνες αξιολόγησης. Ο πρώτος πυλώνας. Εξετάσαμε την στρατηγική συνάφεια και σημασία του blending. Δεύτερος πυλώνας, προστιθέμενη αξία. Και τρίτος πυλώνας, αποτελέσματα των έργων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την στρατηγική συνάφεια, εξετάσαμε το βαθμό στον οποίο ο συνδυασμός ε, δανεισμού ε, και επιχορηγήσεων ήταν σημαντικός ε, στην αρχή της αξιολόγησης, ανάλογα και με τις συγκυρίες σε κάθε χώρα, τις αλλαγές που είχαμε, τις εξελίξεις, αλλά και τις μεταβολές στην ευρωπαϊκή πολιτική και στρατηγική. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το blending επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγαλύτερο βαθμό να επενδύσει και με στρατηγικό πλεονέκτημα, ιδίως ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα οικοδομών μεγάλης κλίμακας και την, την παροχή βοήθειας σε άλλες χώρες ε, για την μετάβασή τους ε, στο καθεστώς γειτονίας. Βοήθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει χώρες που δεν θα ήταν ε, δεν θα μπορούσε να τις ε, προσεγγίσει διαφορετικά. Βρήκαμε ότι στην πλειονότητα των έργων ε, είχαμε να κάνουμε με συγκεκριμένες προκλήσεις που παρεμπόδισαν την υλοποίηση των έργων και έτσι σε πολλές περιπτώσεις το blending χρησιμοποιήθηκε στρατηγικά για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτές τις προκλήσεις και για να πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις ε, στις ε, χώρες εταίρους. Αυτό είναι λοιπόν ένα σημαντικό έβριμα. Ταυτόχρονα η αξιολόγηση δείχνει ότι το blending και πιο συγκεκριμένα για τα πρώτα έργα ε, δεν ολοκλήρωσε, δεν πραγματοποίησε όλες τις δυνατότητές του και δεν αντιμετώπισε τις προκλήσεις των χωρών χαμηλότερου εισοδήματος και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Η αιτιολόγηση ε, της επιχορήγησης δεν ε, τονιζόταν ξανά και ξανά στα πρώτα στάδια της αξιολόγησης. Αυτό τελικά οδήγησε σε μία σειρά έργων που δεν ήταν αρκετά σαφές γιατί χρειαζόμαστε το συγκεκριμένο έργο. Επίσης δεν τονίζαμε συστηματικά το, τους στόχους. Κάποια από τα έργα blending ε, δεν ήταν σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις πολιτικές ε, των χωρών εταίρων, αλλά και με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές σε έναν βαθμό, στο βαθμό που θα περιμέναμε τουλάχιστον. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο βελτίωσης. Και τέλος, δεν υπήρχαν ε, πολλά ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που να συνδέονται. Πάνω το 90% του blending γίνεται ακόμα με τέσσερις βασικούς ε, φορείς. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, KFW, AFD και EBRD. Και η ομάδα εξολόγηση θεωρεί, εξετάζοντα και λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι ε, δεν απερίφθησαν πολλά έργα, θεώρησαν λοιπόν ότι δεν υπήρχε αρκετά υψηλό ανταγωνισμό. Για να έχουμε τελικά τα καλύτερα έργα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προστεθέμενη αξία του blending. Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι το blending σε πολλές περιπτώσεις έχει επιφέρει σημαντική προσταθημένη αξία ε, σε ό,τι αφορά την ε, αναπτυξιακή συνεργασία βάσει επιχορηγήσεων. Υπήρχε μεγάλος αριθμός ε, τέτοιων έργων που έχουν συμβάλει στην προώθηση και τη βελτίωση της πολιτικής στι χώρε εταίρου μέσω και τη τεχνική συνδρομή που έχουμε δώσει πολλά έργα μέσω της επιχορήγησης έχουν οδηγήσει σε εύρωστα έργα που ήταν σημαντικά. Η ομάδα μας αξιολογεί τον σχεδιασμό, την ποιότητα και την τεκμηρίωση των έργων και βρίσκεται τελικά, θεωρεί ότι είναι ε, πολύ ποιοτικά αυτά τα έργα. Και τέλος, οδήγησε στην ενίσχυση του συντονισμού των χορηγών, ιδίω τα πρώτα χρόνια που η εμπλοκή των αντιπροσωπείων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιλογή των ε, έργων ήταν πιο σημαντική. Ταυτόχρονα, για την προσθεθμένη αξία, αξιολόγηση ε, βρήκε και περιπτώσεις, ιδίως για τα παλιότερα έργα και πάλι, Είπα προηγουμένως ότι υπήρξαν περιπτώσεις που υπήρξε και μια θετική επίδραση στις ε, μεταρρυθμίσεις πολιτικής, όμως υπήρχαν και πολλές περιπτώσεις όπου ήταν απογοητευτικά μάλλον τα αποτελέσματα. Το κόστος ε, των συναλλαγών που συνδέεται με τη διαχείριση των έργων ήταν αρκετά υψηλό τελικά. Επειδή το blending έχει να κάνει με μια πλειάδα εταίρων, κάποιες φορές οδήγησε σε περιττές ε, επιπλοκές σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των έργων. Υπήρχε συμμόρφωση με τους κανόνες διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, σχεδόν καθολικά. Η ομάδα λοιπόν βρήκε ότι οι κανόνες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την διαφάνεια τελικά τηρήθηκαν. Όμως η αναγνώριση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν ήταν όσο θα έπρεπε και πάλι συνολικά. Στις συνεντεύξει δηλαδή με τους τελικού δικαιούχου της ε, χώρες εταίρου, δεν υπήρχε επαρκή σύνδεση των έργων ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ομάδα κρίνει ότι σε κάποιε περιπτώσεις αυτό μπορεί να οδήγησε σε απώλεια πολιτικού κεφαλαίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για τον τρίτο πυλώνα που καλύψαμε στην αξιολόγηση, για τα αποτελέσματα δηλαδή των έργων blending, θεωρήσαμε σημαντικό να μην δούμε μόνο κατά πόσο υπάρχει προστιθεμένη αξία από το blending και αν έχουν υλοποιηθεί οι αρχικοί στόχοι, αλλά να εξετάσουμε και τα τελικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέσω του blending και σε τι δηλαδή ακριβώς συμβάλλουμε μέσω των επιχορηγήσεών μας. Και εκεί είδαμε ότι σε μεγάλο βαθμό τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του blending είναι επιτυχή και έχουν ήδη πετύχει τους στόχους τους ή προβλέπουμε ότι θα πετύχουν τους στόχους τους, γιατί κάποια δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Αλλά θεωρούμε ότι βρίσκονται σε καλή τροχιά. Και είναι πολύ πιθανό να πετύχουν τα τελικά, τους τελικούς στόχους και για τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα αποτελέσματα ε, τα απολαμβάνουν τελικοί δικαιούχοι και τα εκτιμούν ιδιαίτερως. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ θετικά. Όμως, η αξιολόγηση δείχνει ότι παρότι ε, σημαντικό στόχο ήταν η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, δεν υπάρχει αρκετή έμφαση στην παρακολούθηση των ε, αποτελεσμάτων των έργων blending σε ό,τι αφορά την δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει καμία επίδραση του blending στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, προφανώ και το κάνει, αλλά δεν έχει ποσοτικοποιηθεί, γιατί δεν το παρακολουθούμε όπω πρέπει και θεωρούμε ότι υπάρχουν και κάποιες ε, χαμένες ευκαιρίες ε, να στοχεύσουμε πιο άμεσα και αποτελεσματικά τους φτωχούς. Υπήρχαν έργα όπου λάβαμε υπόψη την φτώχεια, για παράδειγμα σε ενεργειακά έργα, νομίζω στην Αίγυπτο. Θέλαμε να δώσουμε πρόσβαση ε, σε μία πόλη στην ηλεκτρική ενέργεια και ένα ένας παράγοντας του έργου ήταν να δώσουμε πρόσβαση σε ένα χωριό που ζουν οι πιο φτωχοί. Και έτσι αυτό προσθέθηκε σαν ε, παράμετρος στο έργο για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Έχαμε λοιπόν και τέτοιες περιπτώσεις, όμως συνολικά θεωρήσαμε ότι δεν ε, φτάνουν αυτές οι περιπτώσεις, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτές τις ε, ευκαιρίες. Επίσης, δεν λέμε ότι δεν συμβάλλει το blending στην ε, μείωση της ε, ανέχειας. Ξεκάθαρα αναφέρουμε ότι με τη χρηματοδότηση επιτυχών έργων που έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα, το blending σαφώς και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και βέβαια στο βαθμό που η οικονομική ανάπτυξη είναι συμπεριληπτική, που ξέρουμε ότι δεν συμβαίνει πάντα, μπορούμε εύλογα να αναμένουμε ότι θα έχουμε και σημαντικά ωφέλη και για τους φτωχούς, με έμεσο τρόπο όμως. Εν ώψη και των αδυναμιών που διαπιστώθηκαν, υπάρχουν και μία σειρά συστάσεις στην αξιολόγηση. Να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση ε, στην προσθετικότητα των ε, επιχορηγήσεων blending για να διασφαλίσουμε στο μέλλον ότι για όλα τα έργα θα υπάρχει σαφής και ισχυρή τεκμηρίωση και αιτιολόγηση, ε, να διευρύνουμε τον αριθμό των ε, φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία και έτσι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να έχουμε ψηλότερη ποιότητα έργα να ενισχύσουμε την ευθυγράμμιση των έργων blending με τις εθνικές πολιτικές, όπως είπε προηγουμένως αυτό δεν ίσχυε πάντα, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της ανέχειας και ε, να αυξήσουμε την προβολή όταν αυτά τα έργα είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους ε, πολιτικούς. Αυτά είναι συντομία από πλευρά μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση από τη δική μου πλευρά πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Μιλήσατε γενικά για τη διαδικασία και για τα ζητήματα όλα. Ε, υπάρχει κάπου δημοσιευμένος κατάλογος ε, με τα project έτσι ώστε να ε, έχουμε μια ιδέα ε, ποια είναι τα project τα οποία ακριβώς έχουν δεχτεί αυτήν την κοινή ε, χρηματοδότηση. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ερώτηση, αλλά καλύτερο ο μου να ε, απαντήσει. Ο κύριο Χωσέ Μπαζεμάους, ε, σας δίνω το λόγο αλλά μάλλον καλύτερα πρώτα να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι και μετά να μας πείτε ε, εσείς αυτά που έχετε έτσι ώστε να αποκτήσουμε και εμείς μια καλύτερη αίσθηση σχετικά με το ποια είναι τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζονται, καλύπτονται ας πούμε από, τους, ε, ε, από τα προγράμματα αυτά. Συνάδελφος Κέγγε πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την εισαγωγή ίσως ε, ε, έχω μια ερώτηση η οποία σχετίζεται με αυτό που ρώτησε και η Λίντα. Κάποια στιγμή εσείς αναφερθήκατε στο blending, ε, στην ανάμιξη, ε, που μπορεί να έχει καλό αποτέλεσμα, αντίκτυπο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στην Αφρική το μεγάλο ζήτημα είναι οι νέοι. Κάνατε κάποια έρευνα για να δείτε εάν έχει μέσω του blending ε, βοηθηθεί ε, ή αναπτυχθεί ε, η επιχειρηματικότητα, η έννοια της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων ή των γυναικών. Έχετε βοηθήσει την επιχειρηματικότητα με το blending αυτό. Τα έχετε αξιολογήσει αυτά. Ευχαριστώ. Η Μαρία Χόιποκ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Λίντα. Εσείς ε, είπατε στην έκθεσή σας, στην αναφορά σας τέλος πάντων, ότι μπορέσατε να φτιάξετε γερά έργα στην βάση πολιτικών μεταρρυθμίσεων, επειδή αυτές το επέτρεψαν δηλαδή. Ποιες ήταν αυτές οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις, γιατί συχνά παρατηρούμε ότι γίνονται πολιτικές μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα για αναδασμογιών, που τέλη όμως αποβαίνουν σε βάρος των τοπικών πληθυσμών. Γι' αυτό θα ήθελα να μάθω τι είδου πολιτικές μεταρρυθμίσεις είναι αυτές ε, που, για τις οποίες μιλήσατε. Επίσης με ενδιαφέρει διότι στο τέλος μιλήσατε για προσθετικότητα, additionality. Κατά πόσον έχετε αξιολογήσει εάν οι επενδύσεις αυτές θα γίνονταν και χωρίς την, ε, τον συνδυασμό, το blending δηλαδή. Γίνονται από δημοσίους πόρους. Είτε σπρώχνουμε μια δημόσια χρηματοδότηση και σε έργα τα οποία ούτως ή άλλως θα γίνονταν. Πρόεδρος, πραγματικά η προσθετικότητα είναι πάρα πολύ ε, μεγάλο θέμα. Η κυρία μεγαλο θεμα η κυρια θεοχαρου παρακαλω Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή. Ε, νομίζω ότι το όλο πρόγραμμα έχει τις ίδιες εγγενείς ανομαλίες που έχουν όλα τα προγράμματα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ερώτηση έχω να κάνω. Αν το αξιόχρεο αυτών που θα πάρουν το δανεισμό καλύπτει τις μικρότερες οικονομικά, τις λιγότερο οικονομικά ισχυρές ομάδες των πληθυσμών, διότι αν και πάλι εκμεταλλεύονται το όλο πρόγραμμα οι οικονομικά ισχυροί οι οποίοι θα συνεχίσουν την ίδια προσπάθεια να ξεζουμίζουν τους στόχους καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να γίνει εκείνο το οποίο επιθυμούμε. Και αυτό το ζούμε όχι μόνο στην Αφρική και στις χώρες του τρίτου κόσμου, αλλά και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επειδή δεν έχουν αξιόχρεο οι μικρομεσαίοι, παίρνουν οι μεγάλοι τα κεφάλαια και ε, συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος της ε, μη δημιουργίας θέσεων ή της δημιουργίας θέσεων οι οποίες όμως υποαμείβονται προς όφελος του κεφαλαίου. Ευχαριστώ. Thank you. Lola Ευχαριστώ πολύ, Λόλα Σάντσες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την ε, παρουσίαση. Νομίζω ότι αυτό το blending είναι ε, ε, εύκολο να διαβλέψει κανείς τα προβλήματα τα οποία είναι εγγενή. Υπάρχουν προβλήματα όπως υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν καταδείξει η Oxfam και το ελεγκτικό συνέδριο κτλ. Είναι πολλά τα προβλήματα. Πρώτον, απομακρυνόμαστε από τους βασικούς στόχους, τους αναπτυξιακούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν ασχολούνται με τους πιο ευάλωτους τους ε, ε, ασχολείται και απευθύνεται μονάχα ε, σε χώρες όπου ο επενδυτικός κίνδυνος δεν είναι μεγάλος διότι έχουν ήδη το μέσο εισόδημα. Επίσης είναι πιθανό να μην ευθυγραμμίζονται οι στόχοι του προγράμματος, οι αρχές του προγράμματος με τους στόχους ανάπτυξης και τους στόχους βιωσιμότητας και επίσης δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Αυτά είναι τα προβλήματα του blending. Πιστεύουμε ότι το blending απλώς θέλει να χρησιμοποιήσει ε, την επίσημη ε, ε, βοήθεια, την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια έτσι ώστε να δώσει χρήματα σε κάποιους συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μπορέσει πραγματικά να δώσει λύσεις σε προβλήματα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και τα έχουν καταγγείλει ακόμα και από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου θέλει να πει ο εκπρόσωπο τη ε, Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ για όλα αυτά και μετά θα ξαναμιλήσουμε για την ε, αξιολόγηση. Ναι, βεβαίω μπορώ να προσπαθήσω, κυρία Πρόεδρε, να απαντήσω στα, προβλήματα, στα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν ή μπορεί να αναφερθώ στην ίδια την αξιολόγηση ή μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να συνδυάσετε και τα δύο στοιχεία στην απάντησή σας, λέει η Πρόεδρος. Ίσως λοιπόν καλό θα ήταν να ξεκινήσω με την αξιολόγηση, να σχολιάσω τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Ε, να σας πω λοιπόν ότι ε, το κύριο έβριμα ε, της αξιολόγησης ή μάλλον τα κύρια ευρήματα εμείς τα λαμβάνουμε υπόψη μας ιδιαίτερα σοβαρά και έχουμε και ένα σχέδιο δράσης όπου έχουμε διαπιστώσει ότι οι περισσότερες συστάσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί έχουν ήδη πάρει το δρόμο τους και υλοποιούνται θα προσπαθήσω να μην ε, μακρηγορήσω έτσι ώστε να μπορέσω να απαντήσω και στις ερωτήσεις. Η πρώτη σύσταση αφορά την προσθετικότητα και αυτό είναι κάτι ε, το οποίο μας δυσκολεύει ε, και από την ε, αρχή του προγράμματος. Υπάρχει ένα νέο έντυπο το οποίο ακριβώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι επιδοτήσεις και τα δάνεια. Η προσθετικότητα πραγματικότητα ακριβώς αναφέρεται σε αυτό το ε, έντυπο ε, και ταυτόχρονα αναφέρονται και διάφορα στοιχεία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα, τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία κτλ. Δηλαδή λαμβάνουν, ε, λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία αυτά, αναλύονται στις τεχνικές ε, που γίνονται και εδώ και στα ενδιαφερόμενα κράτη και επομένω ε, γίνεται ενδελεχής ανάλυση όλων αυτών των επιμέρους ε, ε, ζητημάτων. Η δεύτερη σύσταση που προκύπτει από την αξιολόγηση αναφέρεται στην ανάγκη διεύρυνσης των εθνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνεργάζονται μαζί μας σε αυτή τη δραστηριότητα blending. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχουν πολλές περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες οι οποίες συν χρηματοδοτούν τα, τις περισσότερες διαδικασίες. Έχουμε και την Αναπτυξή Γράψα της Αφρικής ε, ε, στα πλαίσια της ε, African Investment Facility. Έχουμε επίσης την ε, τράπεζα, Αναπτυξιακή Τράπεζα της Καραϊβικής ε, για την αντίστοιχη διευκόλυνση. Ε, επίσης έχουμε την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής η οποία συνεργάζεται μαζί μας βεβαίως. Θέλουμε να συμπεριληφθούν και άλλες αναπτυξιακές τράπεζε και για την Νότια Αφρική και για τη Δυτική Αφρική. Έχουμε ήδη ξεκινήσει ε, διαπραγματεύσεις ε, με ε, αυτές τις τράπεζες και προσπαθούμε πραγματικά να παίξουμε σημαντικό ρόλο κατά την έννοια τη συνεργασία μας με τις χώρες αυτές. Επίσης υπάρχουν και διάφορες διευκολύνσεις, facilities οι οποίε μπορούν να συνυπολογιστούν και να παίξουν βέβαια σημαντικό ρόλο. Προκύπτει επίσης και ένα άλλο ζήτημα το οποίο προκύπτει από τις ε, ε, αξιολογήσεις είναι η ευθυγράμμιση με εθνικές πολιτικές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σοβαρότατα λαμβάνουμε υπόψη. Προσπαθούμε να αναλύνουμε τα προγράμματα και σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο και σε όρους πολιτικού συσχετισμού. Ε, γι' αυτό λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη ε, τις ε, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές των εμπλεκομένων. Ιδιαίτερως δεν λαμβάνουμε υπόψη το κατά πόσον υπάρχει εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στη συγκεκριμένη χώρα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι είναι συντονισμένες οι επενδυτικές προσπάθειες. Υπάρχει και άλλη μια σύσταση για διαρκή βελτίωση του σχεδιασμού. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι προς ώρας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί πως ε, ε, η ε, μελέτη η οποία γίνεται και σε πολιτικό και σε επίπεδο στρατηγικής και σε τεχνικό επίπεδο ακριβώς προσπαθεί να διασφαλίσει την, αυτή την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων. Δεν θέλουμε ε, ε, σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε ε, μεγάλη και βαριά γραφειοκρατία. Θέλουμε απλούστευση και εύκολη εκτέλεση. Υπάρχει και μία πραγματική πρόκληση που είναι κάτι που οπωσδήποτε θα προσπαθήσουμε να λύσουμε και με το πρόγραμμα εξωτερικών επενδύσεων είναι το κατά πόσον μπορούμε να εμπλέξουμε ε, περισσότερο την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, κυρίως ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες έγινε και λόγος και πώς ε, θα έχουμε την δυνατότητα να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί κατά αυτήν την έννοια. Όπως έλεγα και προηγουμένως, το γεγονός ότι 1,5 δις έχουν αφιερωθεί ακριβώς ε, για την ε, ε, δημιουργία εγγυήσεων σημαίνει ότι πραγματικά κινούμαστε προς αυτήν την προς αυτήν την οδό και θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε πραγματικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει θυγεί είναι ο αναπτυξιακός αντίκτυπος και η δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω του blending. Ε, αυτό βέβαια ο Άντριαν ήδη το αντιμετώπισε στην αρχική του παρουσίαση. Ωστόσο πιστεύω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι όταν ε, ε, παρουσιάζεται, υποβάλλεται ένα project, οι, τα τέσσερα ιδρύματα, οικονομικά ιδρύματα ε, μας υποβάλλουν και μία εκτίμηση για το πόσες θέσεις εργασίας άμεσες και έμεσες μπορούν να δημιουργηθούν. Επιπροσθέτως δε ε, μας ε, αναφέρουν κατά προσέγγιση τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να ωφεληθούν από το project αυτό. Ανεφέρθη επανειλημμένα το θέμα της Αφρικής και το ανέφερα και εγώ είναι σαφές ότι ο κανονισμός που συζητιέται ε, και αναφέρεται στην πρόταση της Κομισιόν ιδιαιτέρως ε, μεριμνά ε, για την δημιουργία ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Αφρική. Γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στο θέμα αυτό και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην προσπάθεια δημιουργίας προγραμμάτων ακριβώς με αυτόν τον σκοπό, δηλαδή τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Άκουσα μια παρατήρηση και θέλω να σας πω το εξής. Στην αξιολόγηση αναφέρεται ότι σε μερικές περιπτώσεις η διαδικασία προμηθειών στις ε, ε, χώρες δεν είναι ε, αρκετά ευθυγραμμισμένες με τις αρχές της Κομισιόν. Αυτό δεν ισχύει. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε τα καλύτερα δυνατά πρότυπα και όρους και προϋποθέσεις για τις προμήθειες. Τέλος. Το θέμα της ε, ορατότητας. Ε, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι όταν υποβάλλονται ε, τα projects εντό του πλαισίου του blending, η ορατότητα να είναι συγκεκριμένη. Εδώ πρόκειται για μια προσπάθεια κοινή και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της Κομισιόν και των εταίρων. Ζητήσαμε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μας ε, ε, παρέχουν και ένα σχέδιο βιωσιμότητας, το οποίο εξαρτάται κάθε φορά ε, στο project το οποίο υποβάλλεται, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι όσον αφορά την ορατότητα. Αυτά σε σχέση με τις εννέα συστάσεις της αξιολόγησης. Όσον αφορά τώρα τα συγκεκριμένα ερωτήματα, νομίζω ότι ήδη εμέσως απήντησα σε κάποιες από τις ε, ερωτήσεις ε, σχετικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας ε, και είπα ότι ιδιαίτερα για την περίπτωση της Αφρικής αλλά ναι, και μέσω της διευκόλυνσης της γειτονίας αλλά και για την Αφρική γενικότερα οι ε, στόχοι είναι συγκεκριμένοι. Γίνεται δε μέσω των στόχων για την Αφρική και για τη γειτονία μεγάλη εστίαση όσον αφορά την επιχειρηματικότητα των νέων και των γυναικών ιδιαίτερως. Ε, υπήρξε ένα ερώτημα σχετικά με την προσθετικότητα και σχετικά με τις ε, μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι ήδη απήντησα για την προσθετικότητα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, ε, τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε ένα entry point μέσω κυρίως διαλόγου με τον κλάδο, ε, ας πούμε με τον κλάδο της ενέργειας, αυτό είναι το entry point. Με τον τρόπο αυτό ε, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ε, πιο γενικευμένη πολιτική για το περιβάλλον, για την ενέργεια στην χώρα αυτή και ε, με το εργαλείο της ε, γειτονίας για την Αφρική ε, θα μπορέσουμε να βάλουμε, να καταβάλουμε τις προσπάθειές μας από κοινού έτσι ώστε το εργαλείο μας να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικό. Επίσης, ανάγκη μεγαλύτερης εστίασης ε, στην ε, ε, ορατότητα και στην, στις συνέργειες, αυτό το είπα ήδη, θα έχουμε και μια βέβαια μεγαλύτερη εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος, τα πιο κρίσιμα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν προς το τέλος σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι χτες το απόγευμα είχαμε μία συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Κοινωνία των Πολιτών. Ε, είχαμε πάνω από 40 εκπροσώπους ε, στην αίθουσα, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε το External Investment Plan. Μπορώ να σας ε, πω με τα βεβαιότητα ότι ήταν πάρα πολύ καλή η ατμόσφαιρα, ότι οι περισσότερες οργανώσεις ήταν πολύ υποστηρικτικές ε, των προσπαθειών μας ε, ε, και και ήταν όλοι υπέρ ε, του εργαλείου του blending και της δημιουργίας νέου εργαλείου ε, για την γειτονία για την Αφρική. Όσον αφορά ε, τα, τις παρατηρήσεις του Ελληνικού Συνεδρίου, προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Νομίζω και μέσω των, της απάντησης του συστά, στις συστάσεις, άλλωστε, ξεκίνησαμε τη διαδικασία αυτή. Νομίζω ότι ήδη έχουμε προχωρήσει σε κάποιες διορθώσεις και αυτό φαίνεται. Όσον αφορά ότι υποστηρίζουμε περισσότερο τις πιο πλούσιες χώρες. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Εμείς ε, υποστηρίζουμε και χώρες χαμηλού εισοδήματος ε, ε, σε πολλές περιφέρειες δουλεύει το blending όπου έχουμε πιο φτωχές ε, χώρες και μέσω του, σχεδίου, του εξωτερικού σχεδίου ανάπτυξης κάνουμε αυτή την προσπάθεια και τη συνεχίζουμε. Κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουμε κάποια ισορροπία μεταξύ του είδους των χωρών που ωφελούνται από το blending δεν ε, θέλουμε να βοηθήσουμε περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα ε, ή τις ε, χώρες χορηγούς. Υπάρχουν διαδικασίες προμηθειών πολύ συγκεκριμένες και ανοιχτές σε όλους, επομένως δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο όσον αφορά το θέμα αυτό. Να σας πω ότι, ε, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να ευθυγραμμιστούμε με τα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα όσο γίνεται περισσότερο. και να ευθυγραμμιστούμε με αναπτυξιακά προγράμματα εφόσον τέτοια υφίστανται. Μια τελευταία παρατήρηση. Το γεγονός ότι προσπαθούμε να φέρουμε περισσότερους ε, πρωταγωνιστές ε, στο πεδίο της ε, ανάπτυξης σημαίνει ότι απελευθερώνονται και κινητοποιούνται επιπλέον κεφάλαια και επιπλέον πόροι και μάλιστα που θα ευνοήσουν τομείς ε, ε, κοινωνικού, ευρύτερου κοινωνικούς τομείς, την εκπαίδευση κλπ. Α, και κάτι άλλο. Θα δώσω το λόγο, εάν βεβαίω το επιθυμεί, στον Άλγο Μαρτίνς από την Digineer. Γιατί καλύπτονται και οι χώρε τη γειτονία από αυτή την αξιολόγηση. Η Πρόεδρος, αν θέλετε κύριε Μάρτινς, σα δίνω το λόγο. Ναι, για την εφαρμογή των έργων, για την εκτέλεση των έργων. Από την πλευρά ΔΕΦΚΟ υπάρχει μια σελίδα όπου περιλαμβάνονται όλα αυτά τα έργα και περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο. Μέσα στην ίδια σελίδα περιλαμβάνεται και αιτήσια έκθεση για κάθε ένα από το έργο με λεπτομερή περιγραφή του κάθε έργου που εγκρίθηκε για την συγκεκριμένη χρονιά. Άρα όλα τα έργα, όλα τα project και είναι παραπάνω από 300 περιγράφονται καλά μέσα στις εκθέσεις αυτές. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, ακούσαμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχουμε και διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά. Αυτό γιατί, το συμπληρώνω γιατί λυσμόνισε το οποίο Χωσέ. Τώρα, για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, η σεπήρωση των όσων είπε ο Χωσέ, είναι σημαντικό να θυμηθεί κανείς ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι από τους πιο σημαντικούς τομείς για το blending, για ε, την σύζευξη αυτή δανείων με επιχορηγήσεις και ιδίως στις χώρες της γειτονίας έχουμε χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης που διαθέταμε τα τελευταία 2-3 χρόνια για να στηρίξουμε, στηρίξουμε για παράδειγμα συμφωνίες CFDA με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, κάτι που είναι σημαντικό για μας διότι κατευθύνεται απευθείας στην στήριξη της σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών για να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτές τις χώρες οι οποίες θα κληθούν να ανταγωνιστούν με τις ευρωπαϊκές εταιρείες όταν θα ανοίξουν οι αγορές τους. Αυτό είναι ένας από τους τομείς όπου το blending υπήρξε και είναι πολύ χρήσιμο διότι πρόκειται άλλωστε για έργα τα οποία είναι πολύ πρόσφατα Τονίζω δηλαδή ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι από τους μεγαλύτερους τομείς όπου χρησιμοποιείται ε, ο συνδυασμός αυτός. Δεν είναι λοιπόν δίκαιο να πει κάποιος εδώ ότι λησμονούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ένας από τους τομείς όπου στηρίζουμε πολλές επιχειρήσεις αυτές με το blending. Έχετε τίποτε να προσθέσετε? Έγινε μια ερώτηση συγκεκριμένα σχετικά με αυτά που είπα για την συμβολή σε ε, μεταρρυθμίσεις και πώς γίνεται αυτή η συμβολή με το blending. Υπήρξαν περιπτώσεις σε χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφερε και στήριξη του προϋπολογισμού και προσπάθησε μέσω αυτού να περάσει ορισμένες μεταρρυθμίσεις, να προωθήσει ορισμένε μεταρρυθμίσεις σε ορισμένου τομείς και ορισμένα έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν σε ορισμένου τομεί όπου υπήρχαν και policy objectives, υπήρχαν δηλαδή κάποιε περιπτώσει τέτοιε, όπου σημειώθηκε μια συνέργεια ανάμεσα στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του blending και τον διάλογο για τι μεταρρυθμίσεις για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του διαλόγου για τέτοιες μεταρρυθμίσεις σε πολιτικές. Σε ορισμένε περιπτώσει δεν ήταν ακριβώ συστηματική, και υπήρχε και ένας ε, σημαντικός αριθμός ε, περιπτώσεων που δεν συνέβη αυτό. Μάλιστα, μια τελική ερώτηση την οποία απευθύνω ίσως και θέλω να πω ότι τα ζητήματα της προσθετικότητας είναι περίπλοκα. Πριν να γίνω ευρωβουλευτής ε, είχα ασχοληθεί με περιφερειακή ανάπτυξη και με τέτοια θέματα. Τα, ίδια ζητήματα αναφύονται διαρκώς πώς να προχωρήσει ένα συγκεκριμένο project εφόσον δεν έχει δοθεί σχετική χρηματοδότηση. Δουλεύετε με τη Γενική Διεύθυνση Regio που εργάζονται εδώ και δεκαετίες σχετικά και έχουν μηχανισμούς για να μετρούν τις μετακινήσεις των χρηματοδοτήσεων και είναι στάνταρτη οι προσεγγίσεις αυτές για να εξασφαλιστεί τούν τα πιο θετικά αποτελέσματα των επενδύσεων. Επίση, κάτι άλλο που σημειώνουμε όταν κάνουμε αποστολέ στι αυτέ τι χώρε, να ε, ε, κάνουμε πιο συγκεκριμένε ερωτήσει για το blending. Για παράδειγμα, όταν θα πάει η αποστολή μα στο Καμερούν, να ρωτήσει τι γίνεται και στι ενημερώσει που μα κάνουν. Να ρωτήσουμε πιο συγκεκριμένα. όταν έχετε μπροστά σας ένα συγκεκριμένο ε, project, ένα συγκεκριμένο έργο, ε, αποκράτε και μια αίσθηση του τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και πού κατευθύνονται οι ε, χρηματοδοτήσεις. Ευχαριστώ. Είναι εδώ το αφεντικό μου, γι' αυτό διστάζω κάπως να λάβω εγώ το λόγο. Για το ζήτημα της προσθετικότητας πάντως να πω το εξής. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας κυνηγά από την αρχή που αρχίσαμε δηλαδή τις blending activities. Το γεγονός και μόνο ότι δεν έχετε και κάποιο αντίβαρο είναι και δείχνει και πόσο δύσκολο είναι. Πρέπει να λάβετε υπόψη όταν κάνετε μετρήσεις της προσθετικότητας γιατί δεν, ε, εξάλλου βέβαια δεν έχουμε ε, ε, τακτικές ανταλλαγές απόψεων με την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο. Θα το κάνουμε στο μέλλον ίσως. Αλλά να μου επιτρέψετε να σας ε, διαβάσω τα 10 διαφορετικά ζητήματα που περιλαμβάνουν τα δελτία χρηματοδότησης που έχουν σχέση με την προσθετικότητα. Ζητούμε προσθετικότητα δηλαδή για οικονομικούς, χρηματοδοτικούς, κοινωνικούς ε, τομείς, ποιότητα των έργων, βιωσιμότητα, αηφορία, κοινωνική βιωσιμότητα και άλλα σχετικά κριτήρια. Πρόκειται δηλαδή για ένα αριθμό επιχειρημάτων που συμβάλλουν για να αποφασίσουμε τελικά, να κρίνουμε δηλαδή τελικά εάν το συγκεκριμένο έργο είναι εντάσσεται στην προσθετικότητα ή όχι. Πρέπει να απαντηθούν ορισμένε ερωτήσει πρώτα. Ασφαλώς και σας ενθαρρύνουμε να θέτετε ερωτήσεις όταν μεταβαίνετε επιτόπου σχετικά με το συνδυασμό, με το blending. Δεν ξέρω αν εμείς ως Επιτροπή πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Τα τελευταία αυτά χρόνια κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να φτιάξουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει την ποιότητα του έργου, αλλά αυτό μέσα σε βάθος χρόνου. Αρχικά ήταν δύσκολο να πάει κανείς επιτόπου για να δει τι ακριβώς γίνεται με το έργο. Και πράγματι η αξιολόγηση ξεκινά με έργα IPF και LIFE που είναι οι παλαιότεροι μηχανισμοί διευκόλυνσης επενδύσεων και ήταν δύσκολο αρχικά να επιλεχθούν έργα τα οποία να έχουν πραγματική υπόσταση, φυσική υπόσταση και το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασφαλώς θα πρέπει να το λάβουν υπόψη αυτό. Πρόκειται για μεγάλα έργα, δεν μπορούμε να τα ξεκινήσουμε και μετά να τα αφήσουμε στη μοίρα τους. Χρειάζονται παρακολούθηση, υποβολή ξεκάθαρων εκθέσεων και παρακολούθηση για το τι γίνεται από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Και χρειάζεται στενότερη και ισχυρότερη εμπλοκή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδίω από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι επιτόπου. Δηλαδή, ασφαλώς δεχόμαστε τις συστάσεις σας και σας ενθαρρύνουμε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήσασταν σήμερα κοντά μας και ασφαλώς θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά που μάθαμε όταν θα συζητούμε για EFSD. Ευχαριστώ πολύ θα έχουμε τώρα άλλου προσκεκλημένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα εδώ για να μιλήσουν μαζί μας για τη στρατηγική ΑΦΚΟ. colleagues, the e will change the coming. Ε, ε, ε, οι κλητήρε θα αλλάξουν τώρα τι καρτέλε με τα ονόματα μια στιγμή. So, colleagues, we move on now to a very important item. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα ακόμη, το υπαρθμό 18, όπου θα ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο σχετικά με την ανάγκη για νέα όθηση στην εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Η Κομισιόν έχει δημοσιεύσει ανακοίνωση τώρα για την στρατηγική της αυτή στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επόμενη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής που θα γίνει στο Αμπιτζάν τον Νοέμβρη. Θα πάει και δική μας αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στο Αμπιτζάν και θα τα συζητήσουμε βέβαια στα πράγματα αυτά πριν. Μάλιστα σκοπεύουμε να συντάξουμε έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για την στρατηγική για την Αφρική και μάλιστα σήμερα το απόγευμα που θα συναντηθούμε 5 η ώρα θα ορίσουμε και τον σχετικό εισηγητή. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι είναι καλό το ε, χρονικό αυτό πλαίσιο που βρισκόμαστε τώρα για να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πρόκειται να κάνει, τι πρόκειται να αλλάξει και τι μπορούμε να αναμένουμε. Ακούσαμε συχνά την Φεντελίκα Μογκερίνη για το πόσο σημαντική είναι η Αφρική, πόσο μεγάλη είναι η σημασία της Αφρικής. Είναι στο κάτω-κάτω η αυλή μας, αν θέλετε. Και πολύ σημαντικά πράγματα. Μιλήσαμε χθε για τα επίπεδα της ODA, της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, που αυξάνεται η ODA, αλλά το τμήμα της που οδεύει προς την Αφρική μειώνεται. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Όταν μιλάμε για προτεραιότητα, όταν λέμε δηλαδή ότι η Αφρική είναι προτεραιότητα, στην πραγματικότητα βλέπουμε ωστόσο να αυξάνεται το ποσοστό που ε, διοχετεύεται προς Συρία και Ιορδανία. Έχω κοντά μου λοιπόν τον Κουν Ντούνς, Διευθυντή Αρμόδιο για τον Συντονισμό της Ανάπτυξης στην Ανατολική και Μεσημβρή Αφρική, καθώς και τον κύριο Κουν Βερβάκε, διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΙΕΔ για την Αφρική, καθώς και την κυρία Μάρκουσεν, Βρυγκίτε Μάρκουσεν, από Α, και αυτή από την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Ποιο θα ήθελε να αρχίσει πρώτα ο Κούν. Mr. Vavaka, you're going first, because I think yes, it's... Εσείς λοιπόν που εκπροσωπείτε την είπατε εκπρόσωπο. Έχετε το λόγο ευχαρίστω. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε ορισμένες σκέψεις για την προετοιμασία της ε, Συνόδου Κορυφής ε, και περιμένουμε και τη συμβολή της δικής σας Επιτροπής ε, στις εργασίες εν ώψη της Συνόδου. 29 και 30 Νοεμβρίου θα λάβει η χώρα στην Αμπιτζάν. Είναι η πέμπτη ε, μεταξύ των δύο υπήρων και είναι μια σημαντική γιατί έρχεται 10 χρόνια μετά την σύνοδο της Λισαβόνας. Ε, πλέον οι σχέσει μα έχουν μπει σε ε, ισχυρότερες πολιτικές ε, βάσεις και βασιζόμαστε σε, στα κοινά συμφέροντα. Αυτό που τότε αποκαλούσαμε την κοινή στρατηγική μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική. Μια δεκαετία είναι μεγάλο χρονικό διάστημα σε όρου πολιτική και αν ε, δείτε και την στρατηγική του κ. Σολάν αλλά και την στρατηγική παρουσίαση η κ. Ε, Μογκερίνη πέρσι, βλέπουμε τι ε, ευρύτερε προκλήσει που αντιμετωπίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρική και τη σημασία, όπως αναφέρατε και εσείς, της Αφρικής. Για το λόγο αυτό τη στρατηγική δηλαδή σημασία αυτή της σχέσης. Η Αφρική αυτή τη στιγμή περνάει βαθιές και σημαντικές ε, αλλαγές και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο και εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις και για τους δυο μας. Το σημαντικό είναι η Αφρική να πάρει τη θέση της ε, στο διεθνές προσκήνιο και στο Στρασβούρου ακούσαμε τον πρόεδρο μου Μουσαφάκη ε, στην ομιλία του και νομίζω ότι ήταν πολύ ηχηρό το μήνυμά του και με τα χαρά είδα ότι ήταν και θετική υποδοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βλέπουμε λοιπόν και τις αλλαγές από αφρικανικής πλευράς. Από πλευράς μας είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη μας αλλά και εμείς ως ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης συνδέουμε την δική μας ασφάλεια και ευημερία πολύ περισσότερο με τα όσα ε, συμβαίνουν στην Αφρική. Στα τελευταία Συμβούλια Εξωτερικών Υποθέσεων υπήρξαν μακροσκελεί συζητήσει για την Αφρική. Είχαμε μια συζήτηση για το κέρδο τη Αφρικής. τον επόμενο μήνα ε, θα συζητήσουμε για το Σαχέλ. Και βλέπουμε ότι έχει πάρει πλέον πολύ μεγαλύτερη σημασία η Αφρική. Αυτή η σύνοδος κορυφής λοιπόν δεν είναι μία συνηθισμένη σύνοδος. Όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία για να ε, διαμορφώσουμε πραγματική συμμαχία ε, για περισσότερη σταθερότητα και ευημερία. Και αυτό θα έχει θετικά ωφέλη και για τις δύο πλευρές. Υπάρχει μια αίσθηση του επίγοντος που συνδέεται με τις ε, δημογραφικές τάσεις. Όλο αυτό μπορεί να είναι θετικό. Είναι από τις πιο σημαντικές διευθυντικές αλλαγές στον κόσμο και πιο συγκεκριμένα και ιδίως μάλλον στην Αφρική. Όμως υπάρχει και η πρόκληση της απασχόλησης ε, και για το πώς θα δώσουμε ένα μέλλον στα 2,4 ανθρώπους που θα ζουν ε, στην Αφρική σε μερικά χρόνια. Προτείνουμε λοιπόν αυτή η σύνοδος ε, να εξεταστεί υπό το πρίσμα της νεολαίας και αυτό είναι μια θετική διάσταση ενίσχυση της διακυβέρνησης, ε, της ε, χάραξης πολιτικής, ανάπτυξη, απασχόληση, αλλά και παιδεία, μετανάστευση, ρίζοσπαστικοποίηση. Νομίζουμε ότι όλα αυτά αποτελούν ένα καλό σύνολο. Τα όσα παρουσιάσαμε στην κοινή ανακοίνωση περιλαμβάνουν τι αρχικέ μα ε, προτάσει από πλευρά Κομισιόν και τη ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, τα οποία θα συζητήσουμε με την Αφρικανική πλευρά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, θεωρώ. Και σε έναν βαθμό να εξετάσουμε, να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τα κράτη-μέλη μα και έτσι να λάβουμε και τη δική του συμβολή για την ε, υλοποίηση αυτών των προτάσεων. Πρέπει λοιπόν να γίνει ένα κοινό θεματολόγιο που να το οικειοποιούνται και οι δύο πλευρές και να δεσμεύονται προς αυτό. Όμως έχουμε μεριμνήσει ε, να λάβουμε σοβαρά υπόψη και το αφρικανικό θεματολόγιο. Δηλαδή δεν κάνουμε μόνο δικές μας προτάσεις από τις Βρυξέλλες, βασιζόμαστε και στις αφρικανικές ε, προτάσεις ε, με το θεματολόγιο που είχαμε παλαιότερα και το 2017 είναι ένα ειδικό έτος σε ό,τι αφορά τα αφρικανικά ζητήματα και ελπίζουμε ότι οι προτάσει μα θα τύχουν μια ε, θετική υποδοχή από την αφρικανική πλευρά. Βέβαια θα πρέπει να τι ε, εξελίξουμε ε, και να τι αναπτύξουμε περαιτέρω με τις επόμενες εβδομάδες και μήνε. Γενικά έχουμε τρει βασικού στόχου. Πρώτον, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό πάντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξακολουθήσουμε την οικοδόμηση κοινών αξιών και συμφερόντων. Θέλουμε και διμερώς να έρθουμε σε επαφή με όλε τι χώρε, να εμβαθύνουμε το διάλογο, αλλά και συλλογικά με την Ήπειρο και να θέσουμε από κοινού πραγματικά ένα κοινό θεματολόγιο μεταξύ Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική. Ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το είδαμε και στο Παρίσι με την COP21. Το έχουμε αποδείξει και σε άλλε περιστάσει και θέλουμε να το διευρύνουμε αυτό και έτσι να υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό συμμαχία μεταξύ των υπήρων. Δεύτερον, ασφάλεια. Υπάρχει η αντίληψη ότι το να επενδύσουμε στην ασφάλεια στην Αφρική σημαίνει ότι επενδύουμε με αυτόν τον τρόπο και στην ασφάλεια στην Ήπειρό μας και σε χερσαίο και σε θαλάσσιο επίπεδο. Και τρίτον, οικονομική ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε τις θέσεις εργασίας που χρειάζεται η Ήπειρος και αυτό είναι μια ευκαιρία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει, στον ιδιωτικό μας τομέα δηλαδή, να επενδύσει στην Αφρικανική Ήπειρο. Πριν μπούμε στις λεπτομέρειες του πλευρά πολιτικής ασφάλειας και μετά θα δώσω το λόγο στον Κουντούνς, το υψηλό επίπεδο κίνηση σε ό,τι αφορά τη δική μας δέσμευση. Εμείς είμαστε ο πρώτος εταίρο ε, σε ό,τι αφορά την επένδυση, την ανθρωπιστική βοήθεια. Είμαστε ο πρώτος πολιτικός εταίρο και στο εμπόριο, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τη διαφορά αλλά πρέπει και να αναγνωρίσουμε ότι ξεκινούμε ήδη από υψηλό επίπεδο. Και έτσι να εντείνουμε σε ορισμένες περιπτώσεις που χρειαζόμαστε προσαρμογές και όπου πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις. Και σε δύο τομείς θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε σημαντική διαφορά. Πρώτον, πιο ανθεκτικές ε, χώρες, κράτη και κοινωνίες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την ε, ειρήνη, την διακυβέρνηση. Και δεύτερον, το οικονομικό σκέλος, περισσότερε και καλύτερε θέσει απασχόληση και αναπτυξιακό θεματολόγιο. Εν συντομία θα ήθελα να σταθώ στου βασικού τομεί για τον πρώτο κλάδο που ανέφερα, ε, ανθεκτικότητα, αντοχή κοινωνιών και κρατών. Πρώτον, ειρήνη και ασφάλεια. Σε αυτόν τον τομέα ε, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία τα τελευταία δέκα χρόνια, αλλά όπως αναφέρατε, η γειτονία μας πλέον διευρύνεται και ε, συμπεριλαμβάνει και την Αφρική. Από την ε, Βόρεια Αφρική, Δυτική, το Κέρας, αλλά και ακόμα και την Κεντρική Αφρική πλέον. Όλα αυτά μας επηρεάζουν άμεσα. Και η διασύνδεση μεταξύ ε, Λιβύης, μεταξύ του κόλπου και του κέρατος, τη Μεσόγειο, την Κόκκινη Θάλασσα, όλα αυτά απαιτούν την Ερυθρά Θάλασσα. Συγγνώμη, όλα αυτά απαιτούν υψηλότερο επίπεδο δέσμευση με την Αφρικανική Ένωση, αλλά διαφορετική. Που έχουμε αναπτύξει και ε, στην διευκόλυνση για την υποστήριξη προ την Αφρική. Πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούμε σε αυτέ τι νέε προκλήσει. Αυτό έχουμε πρόθεση να κάνουμε και να αναπτύξουμε πολύ ισχυρότερε τριγωνικέ σχέσει μεταξύ Αφρικανική Ένωση, Εθνών και Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε νέα ηγεσία και στον ΟΗΕ και αλλού, οπότε αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Η θαλάσσια ασφάλεια θα αποτελέσει σημαντικό τμήμα. Θέλουμε να στηρίξουμε και την Αφρικανική Ένωση να κινητοποιήσει οικονομικούς πόρους. Θα είναι ένα σημαντικό στόχος. Ξέρετε το σχέδιο Καπερούκα που έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Αφρική. Διακυβέρνηση τώρα. Ήδη είμαστε ο βασικός εταίρος ε, στους διαλόγους μας με την ε, συγκεκριμένη και απτή στήριξή μας ακριβώς όλα αυτά τα ζητήματα της διακυβέρνησης με την τοπική και περιφερειακή διάσταση και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Είναι ένα από τα κύρια ζητήματα της σχέσης μας. Η διακυβέρνηση είναι θεμελιώδης σημασία για την σταθερότητα Επομένω, ε, σε αυτό συμφωνούμε. Έχουμε κοινέ αξίε, αλλά πρέπει να δούμε πώ όλα αυτά θα υλοποιηθούν στην πράξη. Και αυτό θα εξετάσουμε με του Αφρικανού εταίρου μα, γιατί ξέρουμε ότι και η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσει σε αυτό το επίπεδο. Και θέλουμε ιδίω να επικεντρωθούμε στην εκλογική διαδικασία. Δημοκρατία, διακυβέρνηση, όπου τα τελευταία χρόνια είδαμε οι παρατηρητές δηλαδή στην εκλογική διαδικασία βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, διαφωνίε μεταξύ Αφρική και Ευρωπαϊκής Ένωση. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού μπορούμε να εμβαθύνουμε και να προωθήσουμε αυτό το θεματολόγιο. Τέλος, μεταναστεύση και κινητικότητα. Δεν θέλουμε αυτή η σύνοδος να αφορά μόνο τη μετανάστευση, Όμω, για πολλά από τα κράτη-μέλη μα, σίγουρα θα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα συζητηθεί. Όμως θέλουμε να συζητηθεί και στο πλαίσιο ενός ε, υπηρετικού θεματολογίου. Μόνο μια μικρή μειοψηφία ε, της μετανάστευσης φτάνει ε, στην Ευρώπη. Το 90% των μεταναστών κινείται εντός της Αφρικανικής Επίρου και πολλές χώρες της Αφρικής αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που, που αντιμετωπίζουμε και εμείς, της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Πρέπει λοιπόν να έχουμε το κατάλληλο ε, θεσμικό πλαίσιο, ούτως ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις στην Ήπειρο. Αυτό είναι ένας στόχος μας και θέλουν τη συνεργασία μας και τη στήριξή μας. Η ε, εμπορία ανθρώπων είναι μια πρόκληση και στην Αφρική και έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ε, πλαίσιο, έχουμε πλέον ε, εμπειρογνωμοσύνη και μέσω της διαδικασίας της Βαλέτας και έτσι μπορούμε όλα αυτά να τα διευρύνουμε περαιτέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Κουν νούμερο 2 τώρα. Ευχαριστώ. Να συνεχίσω αυτά που είπε ο Κούν. Ε, παρουσίασε τις δύο βασικές ε, πλευρές δράσης, ανθεκτικά κράτη. Σε αυτό στάθηκε εκείνο περισσότερο. Εγώ θα ε, επεκταθώ περισσότερο στο δεύτερο σκέλος, την απασχόληση. Θέσεις εργασίας, ιδίως για την νεολαία και για τις γυναίκες. Το εργασιακό θεματολόγιο είναι κέρια γιατί θα πρέπει να το εξετάσουμε και στο πλαίσιο των δημογραφικών τάσεων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ξανά και ξανά εγείρεται κάθε φορά που μιλούμε με τους ε, Αφρικανούς εταίρους μας, είτε σε εθνικό, σε τοπικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Η ανακοίνωση παρουσιάζει ουσιαστικά τέσσερις βασικούς γνώμονες δράσεις υπό το κεφάλαιο της απασχόλησης. Πρώτον, προσέλκυση επενδύσεων. Αν δείτε ε, το ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης ε, στην Αφρική τα τελευταία δέκα χρόνια, βλέπουμε ότι τα στοιχεία είναι καλά, είναι εντυπωσιακά ε, εκ πρώτης όψεως, αλλά αν τα εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος, τα περισσότερα αφορούν εξάρτηση από εμπορεύματα, εξαγωγή πρώτων υλών, ε, βασιζόμενοι στην κινέζικη ανάπτυξη. Όμως, ε, η πραγματική δυναμική έγκυται στην προσθήκη αξίας. Οι δυνατότητες υπάρχουν, αλλά απαιτούνται επενδύσεις για να πραγματοθούν όλα αυτά. Η πρώτη προτεραιότητα λοιπόν, και ξέρω ότι έχετε ε, εξετάσει ακριβώς πριν στο σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων, είναι να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα να ρέουν προς την Αφρική, περισσότερες κεφαλαιακές επενδύσεις από ό,τι σήμερα. Έχουμε λοιπόν ε, τις δυνατότητες, αλλά δεν ε, υλοποιούνται ακόμα στο έπακρον. Το Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Σχέδιο Επενδύσεων είναι μια προσπάθεια διευκόλυνσης αυτής της διαδικασίας μέσω της, ε, του, του δανειστικού σκέλους και μέσω της διευκόλυνσης ε, για τις ε, εγγυήσει και στον δεύτερο πυλώνα για την συνδρομή και για το σκέλος που αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα θέλουμε να διαμορφώσουμε καλύτερο πλαίσιο για τις ε, σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Έχουμε διαμορφώσει μια πλατφόρμα όπου μπορούν ε, μέσω της οποίας να συνομιλούν οι επιχειρήσεις και βλέπουμε ότι αυτό είναι θετικό. Τρίτον, Θέλουμε να βοηθήσουμε ε, στην οικοδόμηση περιφερειακών αγορών περισσότερο από τη σήμερα. Αν θέλουμε προστιθέμενη αξία και επενδύσεις, προφανώς και χρειαζόμαστε πελάτες για τα προϊόντα. Πολλές από τις εθνικές αρχές αγορές είναι πολύ μικρές. Γι' αυτό και θα πρέπει να δημιουργηθούν περιφερειακές αγορές. Υπάρχει ένα θεματολόγιο περιφερειακή ολοκλήρωση στην Αφρική. Είναι δύσκολο βέβαια, έχει προκλήσει. Εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους Αφρικανούς εταίρους μας να πετύχουν και ε, να υλοποιήσουν το ε, θεματολόγιο περιφερειακής ολοκλήρωσης. Ε, για παράδειγμα, έχουμε την τριμερή συμφωνία που συνδέει επιμέρους περιφέρειες και βέβαια στήριξη και για την υπηρετική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Όλα αυτά είναι ένας τρόπος ε, να βοηθήσουμε τους εταίρους μας να υποφεληθούν στο έπακρον των οικονομικών συμφωνιών, γιατί βασίζεται στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας ε, και στην δημιουργία των παραγωγή προϊόντων από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος λοιπόν, συνδέεται με την ε, οικονομία προστιθέμενης αξίας, επηρεάζουμε δηλαδή την ελκυστικότητα για τις επενδύσεις. Δεύτερον, δίνουμε έμφαση σε δύο πιο συγκεκριμένου τομεί ε, και κλάδου όπου απαιτούνται πραγματικέ προσπάθειε. Ο πρώτο είναι ο τομέα τη ενέργεια και πιο συγκεκριμένα τη ανανεώσιμη ενέργεια. Είναι θεμελιώδη σημασία γιατί η ενέργεια είναι κλειδί για πολλούς από τους στόχους μας, όχι μόνο για τι επενδύσει. Προφανώ χωρί την ενέργεια δεν έχουμε επενδύσει. αλλά και για την παροχή βασικών υπηρεσιών. Και στο δίκτυο και εκτός. Σε πολλά, σε πολλά μέρη υπάρχουν ε, προοπτικές και δυνατότητες, ιδίως για τα φωτοβολταϊκά, τεράστιες ε, δυνατότητες. Ένα ε, φωτοβολταϊκό πάνελ παράγει την διπλάσια ενέργεια στην Αφρική από ό,τι στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν έχουμε όλα τα φόντα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Έχουν το δικό τους θεματολόγιο, το οποίο είναι βασικό στοιχείο για εκείνου ε, για την ε, υλοποίηση των στόχων τους ε, για την COP21 και εδώ α πούμε πραγματική πίεση κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τους Αφρικανούς εταίρου μας να υλοποιήσουν τους στόχου. Ξέρετε και Μίμητσα ε, είναι και μέλος ε, του ε, Διευθυντικού Συμβουλίου του ΑΡΕΙ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν με την Αναταξιακή Τράπεζα για να βοηθήσουμε. Βέβαια δεν είναι μόνο θέμα αυτών των μεγάλων έργων. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις και την διακυβέρνηση σε επίπεδο δήμων ή περιφερειακή συνεργασία σε ό,τι αφορά την έρευνα. Τρίτος τομέας. Γεωργία και Αλία. Σαφώς και η γεωργία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην Αφρική για πολλούς λόγους. Ε, απασχολεί το μεγαλύτερο τμήμα ε, του πληθυσμού, ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό από πλευρά σύντησης του πληθυσμού, αλλά δεν έχουμε και πραγματικές δυνατότητες ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Εντάξει, δεν μπορώ να, μιλήσω ακριβώ για αγροεπιχειρηματικότητα, γιατί αυτό μας δίνει την εικόνα ότι έχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο, αλλά αν δούμε τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες, μπορούμε χωρίς πολύ μεγάλες επενδύσεις να βοηθήσουμε τους μικρούς γεωργούς να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους, να τους φέρουμε σε επαφή με αγορές, να τους ενημερώσουμε για την αξία του προϊόντος τους, να τους συνδέσουμε με την τοπική εθνική αγορά και εδώ έχουμε πραγματικές δυνατότητες που ταυτόχρονα ε, βοηθούν τον κόσμο να ξεφύγει από τη φτώχεια, τους ε, παρέχει πραγματική προοπτική και ταυτόχρονα παρέχει και προσταθέμενη αξία σε σχέση με τα όσα παράγονται αυτή τη στιγμή. Ε, αντίστοιχο είναι και το εγχείρημα για την αλληλεία. Όλος ο κλάδος της αλληλείας, της παράκτιας ανάπτυξης, έχει τεράστιες δυνατότητες που αυτή τη στιγμή υποτιμάται και δεν αναπτύσσεται όσο πρέπει. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος στο οποίο θέλουμε να επικεντρωθούμε. Με όλα αυτά συνδέονται βεβαίως και η κατάρτιση με βάση τις δεξιότητες και η έρευνα. Ανάπτυξη λοιπόν δεξιοτήτων μέσω της ε, επαγγελματικής ε, κατάρτισης τεχνικής και δεύτερον έρευνα θέλουμε να κάνουμε περισσότερα παρότι κάνουμε ήδη πολλά Ιδίω για να στοχεύσουμε και να κατευθύνουμε την έρευνα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ωφεληθούν οι Αφρικανοί εταίροι. Τέλος, ε, δεξιότητες. Όλα αυτά δεν έχουν νόημα αν δεν επενδύσουμε ε, στους πολίτες και στην κατάρτισή τους. Επομένως, ε, εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα με ειδική εστίαση στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση και με ιδιαίτερη έμφαση ε, στο Erasmus Plus και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ως ε, σημείο κίνησης και να διαβρύνουμε τις ε, σχέσεις μας με την Αφρική. Θα μείνω εδώ. Όλα αυτά βέβαια δεν αντικατοπτρίζουν όλο το φάσμα της αναπτυξιακής μας πολιτικής και τις σχέσεις μας με την Αφρική. Είναι Έχουμε ένα κάτι πολύ πιο διευρυμένο από αυτό που σας παρουσιάζουμε τώρα. Η ανακοίνωση λοιπόν δεν αντανακλά το σύνολο των σχέσεών μας με την Αφρική. Όπως είπε και ο Κούν, ο σκοπός είναι πολιτικός. Ο σκοπός είναι πολιτικός. Θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε ένα ε, κέντρο βαρύτητας γύρω από το οποίο μπορούμε να εργαστούμε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής και μετά τη Σύνοδο. Μία από τις βασικές προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας είναι αυτή. Όπως είπε και ο Κούν, και δεν το αναγνωρίζουμε πάντα, αν διαβάστε άρθρα για την Κίνα, για την Ιαπωνία, εμείς είμαστε ο υπαριθμόν ένα εταίρος της Αφρικής. Νούμερο ένα πάροχος ε, άμεσης βοήθειας, βοήθεια, βοήθειας, ε, εμβασμάτων και πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος. Θέλουμε να κάνουμε βέβαια περισσότερα. Αν δείτε λοιπόν τα στοιχεία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Όμως, κατά κάποιο τρόπο και πάλι, πάντα πάμε εκεί λίγο αποσυντονισμένοι. Θέλουμε λοιπόν τώρα, και αυτός θα είναι και ο στόχος των συζητήσεων στο Συμβούλιο, να πάμε στην Αμπιτζάν όχι μόνο με τα όσα παρουσιάζουμε ως Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά με πραγματικό ενιαίο θεματολόγιο, που θα περιλαμβάνει τα όσα κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη μας διμερώς. Εάν δεν τα καταφέρουμε να δείξουμε όσα κάνουμε ήδη ε, και τα όσα θέλουμε ακόμα να πετύχουμε, πάντα θα προβάλλουμε μια εικόνα που μας αδικεί ε, σε σχέση με τα όσα μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα στοιχείο ομοσπονδιοποίηση του θεματολογίου εντό εισαγωγικών. Ε, αυτό είναι ένα στόχος της ανακοίνωση. Θέλουμε σε κάποια σημεία, όχι σε όλα, αλλά σε κάποια θα πρέπει να επικεντρωθούμε και ε, να κινητοποιηθούμε από κοινού. Και έτσι, με μεγάλη προσμονή, περιμένουμε και τη δική σας ε, συμβολή μέσω της ε, δικής σας ε, πρωτοβουλία, ε, συγγνώμη, έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας σίγουρα θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ εσείς κύριε Μάκενσον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα να επεκταθώ λίγο σχετικά με το μορφότυπο. Θέλουμε καινοτομία και συμπερίληψη των νέων. Το βασικό θέμα μας είναι οι νέοι, η νεολαία. Θέλουμε όμως και να φτιάξουμε μια διαδικασία που θα προσελκύσει τους νέους να εμπλακούν και βλέπουμε και ορισμένους νεο, νεαρούς Ευρωπαίους και νεαρές Ευρωπαίες στο βάθος της αίθουσας και μιας και μιλούμε για νεολαία, πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Θέλουμε λοιπόν τέσσερα βήματα που έχουμε, δηλαδή έναν αριθμό συναντήσεων και έναν αριθμό ε, βημάτων σχεδιασμού με συμμετοχή νέων από την Ευρώπη και νέων από την Αφρική. Σε ένα δεύτερο βήμα θα γίνει ένα φόρουμ νεολαίας τον Σεπτέμβρη και μετά από αυτό το φόρουμ νεολαίας θα κάνουμε δύο προπαρασκευαστικές διασκέψεις. Το ένα θα λέγεται plot in φάση με συμμετοχή πάλι νέων από την Ευρώπη και την Αφρική για να ε, προχωρήσουν σιγά σιγά μέχρι την πραγματική διάσκεψη κορυφής όπου θα έχουμε σημαντική, σημαντικές εισρωές από τους νέους και τις νέες και για τη διάσκεψη κορυφής. Αυτό ήθελα να πω λοιπόν με λίγα λόγια, διότι αυτό είναι σημαντικό. Θα πρόκειται για, μια διαφορετική διάσκεψη κορυφής αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος και εγώ για την πραγματικά πολύ συνεκτική ε, ε, άποψή σας. Αρχίζω και αντιλαμβάνομαι περί τίνος πρόκειται και αντιλαμβάνομαι και περί τίνος δεν πρόκειται διότι η σύγχυση όταν μιλούμε για το μέλλον της εταιρική σχέσης, μιλούμε για περιφερειακές λωρίδες μέσα στην ίδια την εταιρική σχέση, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν μιλούμε για ολόκληρη στρατηγική για την Αφρική, αλλά να δοθεί μια πολιτική όθηση ξανά στην απομακρού χρόνου ε, εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Charles Goerens. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις ομιλητές ε, της ε, Κομισιόν και του, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Όταν γνωρίζει κανείς λίγο πώς γίνονται αυτές οι διεθνείς ε, διασκέψεις κορυφής, ε, κατανοεί και γνωρίζει ότι ε, δεν αποφασίζονται και πολλά πράγματα έως και τίποτα ε, στη διάρκεια του ίδιου του ΣΟΜΕ, της ίδιας διάστασης κορυφής, αλλά δεν αποφασίζονται πράγματα εκείνη τη μέρα ή πολύ σπάνια. Αλλά το σημαντικό είναι τι γίνεται μετά, πώς είναι δυνατόν δηλαδή να διαμορφωθούν εταιρικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μειώσω την σημασία αυτής της διάσκεψης κορυφής ε, προς Θεού. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια δυναμική αλλαγή. Ε, υπάρχουν κάποιες τέτοιες, ε, κάποιες τέτοιες ενδείξεις που βάζουν λοιπόν τη σχέση μας με την Αφρική σε μια άλλη διάσταση. Έχουμε 5% ας πούμε ανάπτυξη στην Ιγυρία. Ωστόσο, Ωστόσο, πρέπει να αφαιρέσουμε τρία, ε, τρεις ε, ποσοστιαίες μονάδες, ε, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δημογραφική αύξηση. Πρέπει, επομένως, το θέμα το δημογραφικό να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει, επίσης, η τρομοκρατική απειλή. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί οπωσδήποτε μεγάλη αστάθεια. Δεν ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, ωστόσο γνωρίζουμε ότι θα διαρκέσει ακόμα για πολύ και ότι οπωσδήποτε ε, θα ε, χρειαστεί για την αντιμετώπιση του πόρους τους οποίους οι αφρικανικές χώρες δεν έχουν, δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή. Επίσης, ε, το θέμα της ανάπτυξης υπάρχουν χώρες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιο πλούτο και μπορούν, εάν θελήσουν βεβαίως, να ανακατανείμουν ένα μέρος αυτού του πλούτου σε άλλες χώρες. Απαντώντα ε, και στι ε, απαιτήσει των στόχων βιώσιμη ανάπτυξης. Και έπειτα υπάρχει και ένα περίεργο φαινόμενο που ε, αφορά την στασιμότητα ή ακόμα και οπισθοχώρηση των τιμών των πρώτων υλών. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρώπη έχει δυνατότητες πλέον να είναι πλέον παρούσα και να είναι πλέον ορατή και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί όντω μεγάλη ορατότητα σε αυτή τη σχεση Αφρική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχει όμω και ένα σκόπελο που πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί. Υπάρχουν διάφορε σχέσει ε, συνεργασίες, ε, οι οποίε μπορεί να είναι οικονομικέ, μπορεί να αφορούν την ασφάλεια, πάρα πολύ ωραία ε, και βεβαίω θα πρέπει να γίνει και ένα κατάλογο των ενδιαφερόντων από με τη μία πλευρά και από την άλλη, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει όμω και μία επικεφαλή να ε, ανάπτυξη σε όλα αυτά. Και υπάρχει και η υποχρέωση της ε, ε, άμεσης και ανεξάρτητης βοήθειας και επομένως δεν θα πρέπει, δεν θα πρέπει όλες αυτές οι προσπάθειες να περνούν μέσα από, την αναπτυξιακή, από το εργαλείο της αναπτυξιακής βοήθειας γιατί θα αποτύχουν αυτές οι προσπάθειες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από, την άποψη της ανάπτυξης ε, θα πρέπει ε, να δούμε ένα φαινόμενο το οποίο ακόμα δεν κατέχουμε και καλά. Μήπως σε αυτήν τη διάσκεψη θα μπορούσαμε να μελετήσουμε το κατά πόσο η Αφρική μπορεί να έχει μια αναπτυξιακή ε, πορεία παρόμοια με τις, αυτήν τη Λατινικής Αμερικής, πολύ πλούσιοι, πολύ φτωχοί, λίγοι στη μέση τάξη και πολλές απειλές. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να οργανώσουμε καλά την, την εταιρική σχέση. Θα πρέπει να πείσουμε τους Αφρικανούς να εμπλακούν σε αυτή τη συζήτηση, γιατί αν δεν το θελήσουν δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε. Ε, μπορούν να μας πούνε, ε, έχετε κι εσείς ήδη πολλά προβλήματα ή και εμείς έχουμε πολλά προβλήματα ε, στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τις ανισότητες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι γι' αυτό. Ε, μπορούμε να βρούμε ας πούμε ε, το θέμα της, να δούμε το θέμα της ε, φορολογίας. Είπατε κι εσείς, τα θέματα της διακυβέρνησης είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα κοινωνικά επίσης. Μπορώ να σκεφτώ λίγο τι μέσα διαθέτουμε, ας πούμε. Έχουμε το, ταμείο, ε, το αναπτυξιακό ταμείο. <coughs> Μπορούμε να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε κάποιους μεγάλους άξονες ε, και όχι να προσπαθήσουμε να κάνουμε πολλά, υπερβολικά πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Στη Ρουάντα, ας πούμε, πάνω από 80% των ε, ε, κατοίκων, των πολιτών, έχουν πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση. Το Μαλάουι δεν ε, προχωράει τόσο καλά, δεν πάει τόσο καλά οικονομικά, αλλά παρόλα αυτά ε, έχει δώσει πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση στους περισσότερους πολίτες. Επομένως, ακόμα και μια χώρα όπως το Μαλάουι, με προφίλ τελείως διαφορετικό, εκ διαμέτρου αντίθετο από τη Ρουάντα, μπορεί να λειτουργήσει καλά σε έναν ε, ε τομέα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε πολλά μέσα, αποτελεσματικά μέσα για την ε, ανακατανομή του πλούτου. Και, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για βέλτιστους τρόπους παρέμβασης ή ε, κίνησης. Ε, ναι, βεβαίως, είναι πολύ σημαντική η συνεργασία που ε, ανακοινώσατε. Αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει παραπέρα η οικονομική συνεργασία σε πλαίσια ανάπτυξης έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε να εκριζώσουμε την φτώχεια όμως αντιμετωπίζοντας τους αναπτυξιακούς στόχους με κοινούς όρους. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της Αφρικής. Πολύ τροφή για σκέψη, ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Χόιμπουχ. Α, εσείς θα προσθέσετε και άλλη τροφή για σκέψη. Ναι, θα μιλήσω και εγώ μάλιστα για ωραίες μαγειρικές συνταγές. Ευχαριστώ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις που δώσατε. Κύριε Βεράικεν, μιλήσατε πολύ για ασφάλεια, για σταθερότητα. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες αμφιβολίες. Ασφαλώ, η ασφάλεια είναι σημαντική και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων. Οι δικέ μου αμφιβολίε έχουν ω εξή. Πώς χρηματοδοτούνται και από πού μέτρα για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Οι δικέ μου αμφιβολίε είναι ότι εάν όλο και περισσότερο, και αυτό παρατηρούμε, παίρνουμε χρήματα από την αναπτυξιακή πολιτική για να χρηματοδοτούμε τέτοια πράγματα, τότε μας λείπουν τα χρήματα για αυτά που λέει ο άλλος συναδελφός σας, που μιλεί για ανάπτυξη, για απασχόληση. Jobs, jobs, jobs. Το πρόβλημα της ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπιστεί με κατάλληλους μηχανισμούς, να χρηματοδοτηθεί δηλαδή με κατάλληλους μηχανισμούς και όχι από τους πόρους της αναπτυξιακής πολιτικής. Αυτή είναι η πρώτη αμφιβολία που έχω να σας εκθέσω. Μετά μιλείτε για επενδύσεις, περισσότερη ντόπια μεταποίηση για να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση όπου τα έσοδά τους είναι μονάχα από εξαγωγές πρώτων υλών. Το προσυπογράφουμε αυτό. Χρειάζεται περισσότερη μεταποίηση επιτόπου. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη τότε, επειδή άπαξ γίνεται η μεταποίηση των πρώτων υλών, θα χρειαστεί εμείς να αποδώσουμε ένα τμήμα της μεταποίησης. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την τόφια μεταποίηση, δεν θα γίνεται πλέον η μεταποίηση παροιμήν. Είπατε επίσης δημιουργία περιφερειακών αγορών. Όντω αυτό θα αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη λογική συνέπεια. Δηλαδή γίνεται επιτόπου η μεταποίηση, άρα διοχετεύονται και τα προϊόντα επιτόπου. Άρα οι άνθρωποι μπορούν και να αγοράζουν τα προϊόντα που παράγονται επιτόπου σύμφωνοι. Ε, Επομένω αυτό οδηγεί στη δημιουργία περιφερικής αγοράς. Αλλά κάποια ανησυχία έχω ως προς το εξής. Στο ίδιο πλαίσιο είπατε ώστε να μπορούν να υποφελούνται περισσότερο από τα μέτρα έπας οι χώρες αυτές. Καμιά φορά με ανησυχεί όταν εξετάζουμε τι γίνεται στην Αφρική ότι προσπαθεί η Αφρική να δημιουργεί τοπικές αγορές, για παράδειγμα οι χώρες της Ανατολικής Αφρικής, προσπαθούν να φτιάξουν εκεί ζώνες ελευθέρων συναλλαγών, να φτιάξουν ένα είδος αφρικανικής ενίας αγοράς, όπως έχουμε εμείς εδώ την Ευρωπαϊκή. Κατά πόσο τα μέτρα ΕΠΑΣ το υπονομεύουν αυτό, υπονομεύουν την προσπάθεια αυτή, διότι μπορεί εν τέλει να είναι και ελκυστικότερο να φτάσει ένα προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά που θα πολιθεί σε υψηλότερη τιμή, και να μην μείνει σε αυτή την τόπια αφρικανική εντό εισαγωγικών έννοια αγορά. Άρα μπορεί να αναπτυχθεί κάποια κατάσταση ανταγωνισμού. Θα πρέπει να προσέξουμε να του αφήσουμε εκεί το αναγκαίο περιθώριο ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν περιφερειακές αγορές. Τέλος, για την γεωργία. Συμφωνώ μαζί σας ότι στην Γεωργία υπάρχει μεγάλο δυναμικό στην Αφρική. Αφενός μεγάλο δυναμικό, διότι οι άνθρωποι πεινούν εκεί. Άρα πρόκειται για μεγάλη αγορά η οποία υφίσταται. Εξάλλου υπάρχει και μεγαλύτερο δυναμικό παραγωγής. Μόνο να μην κάνουμε το σφάλμα, να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε και να επιβάλλουμε τις παραγωγικές μας μεθόδους που οδηγούν, ως γνωρίζετε εδώ στην Ευρώπη, σε μια μεγαλύτερη εκβιομηχάνηση της γεωργίας. Έχουμε προβλήματα εδώ στην ε, Ευρώπη. Εγώ είμαι μάλιστα αγρότησα και γνωρίζω για ποιο πράγμα σας μιλώ. Φτάνουμε στα όρια της εκβιομηχάνησης. Και θα φτάσουμε πολύ σύντομα. Παρόλο που εδώ έχουμε πραγματικά πολύ καλές προϋποθέσεις για τη γεωργική παραγωγή, που συχνά αυτές οι συνθήκες που εδώ είναι ευνοϊκές δεν είναι καθόλου δεδομένες στην Αφρική. Το δυναμικό λοιπόν μεγαλύτερη παραγωγή θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στην Αφρική, αλλά με διαφορετικέ μεθόδου. Μιλήσατε για έρευνα. Σωστό. Πρέπει να αναπτυχθεί έρευνα. Να αναπτυχθούν μέθοδοι οικολογικέ γεωρική παραγωγή. Αυτό θα είναι όσο, όλο και πιο σημαντικό, διότι δεν αρκεί το λίπασμα, χρειάζεται και νερό. Το νερό δεν υπάρχει παντού απεριόριστο. Θα χρειαστεί λοιπόν να αναπτυχθούν μέτρα για να αυξήσουν και την απορροφητικότητα του εδάφους για το νερό. Αγροτικές λοιπόν οικολογικές μέθοδοι, ασφαλώς χρειάζεται και πολύ επαγγελματική κατάρτιση, να μην κάνουμε όμως ξαναλέω το σφάλμα να προσπαθήσουμε να εξαγάγουμε τις δικές μας εκφιομηχανισμένες μεθόδους γεωρικής παραγωγής. Ότι δηλαδή, να νομίζουμε δηλαδή ότι α, αν ρίξουμε περισσότερο λίπασμα, περισσότερα μηχανήματα κτλ. θα αυξηθεί και η παραγωγή. Σήμερα το πρωί συμμετείχα σε πρόγευμα με μια μη κρατική οργάνωση που λέγεται Ψωμί για τον κόσμο και μια εκπρόσωπος από την Αργεντινή όπου και εκεί έχουν παρόμοιες συνθήκες λίγο με την Αφρική και μας και γράψει εκεί ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν εκεί τώρα τα οποία προέκυψαν από αυτού του είδους την Γεωργία. Όλα αυτά τα σφάλματα δεν επιτρέπεται να τα επαναλάβουμε στην Αφρική. Δυστυχώ τώρα οφείλω να αποχωρήσω γιατί ε, είμαι υποχρεωμένη να πάω σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή και δεν θα μπορέσω να ακούσω τι απαντήσει σα, αλλά θα μου τι μεταφέρουν. Να έρθω σε ορισμένα ζητήματα που έθεσαν οι συναδελφοί μου. Πρώτα του Σαλ Γκέρετ που λέει σωστά ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και υπάρχει δυνατότητα ορισμένε αφρικανικέ χώρε να δείξουν ηγετική ικανότητα και να αποτελέσουν πόλους έλξης. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό ένα είδος κράτους κοινωνικής ευημερίας. Ο Μπαν Κιμούν μίλησε για αυτό σε ένα από τους τελευταίους λόγους που, εξεφώνησε πριν να αποχωρήσει από τα Ηνωμένα Έθνη και ένα είδος universal health care εμείς φτιάξαμε τα κράτη κοινωνικής ευημερίας όταν, όχι όταν είχαμε ε, οικονομική ευημερία, αλλά ακριβώς αμέσως μετά τον πόλεμο, σε δύσκολες συνθήκες. Και οι υπηρεσίες υγείας φτιάχτηκαν στη χώρα μου το 1947, μέσα σε βαθύτατη οικονομική κρίση. Όμως υπήρχε η πολιτική όθηση για να γίνει κάτι. Και είχαμε και την ελπίδα για το μέλλον, θα αλλάξει η ζωή και δεν θα είμαστε πλέον μόνοι μας. Οι πολίτες δηλαδή. Ίσως μπορούν να εμπνευστούν από ορισμένα καλά παραδείγματα. Πριν από δύο χρόνια είχα πάει σε μια ε, διάσκεψη που λιγόταν γυναίκες στα κοινοβούλια και συζητήσαμε εκεί για βασικά ε, συστήματα, μάλλον κοινωνικής ευημερία και ασφάλειας. Καλύτερα τέτοια πράγματα παρά να μιλούμε με λόγια του αέρα για επενδύσεις, απασχολήσεις και ούτω καθεξής. Αυτά θα οδηγήσουν, αυτά θα δώσουν κάποιες λύσεις στους νέους. Δεν υπάρχουν ε, θαυματουργές λύσεις. Και όταν βλέπω και τι γίνεται στην Ισπανία, στην Ελλάδα και αλλού που έχουμε πάρα πολύ υψηλή ανεργία νέων, με απασχολούν και αυτά. Με αυτά θα δώσουμε ελπίδα στον κόσμο. Γιατί ξέρω ότι και η Μαργαρίτα, ε, και η κυρία Μογκερίνη μάλλον, ε, μίλησε την ανάγκη να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο. Και είπατε ότι η Ευρώπη είναι σημαντική και έχει μεγάλη επιρροή στην Αφρική. Ποια θα είναι η συνέπεια της Βρετανικής εξόδου. Αφρικανοί πρέσβεις με ρωτούν αν θα εξαφανιστεί το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί είναι σημαντικός παίκτη στην Αφρική το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ο Σάλ ρώτησε τι θα γίνει με το Brexit και μας απασχολεί και μας. Πώς το βλέπετε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει η Βρετανική κυβέρνηση στο μέλλον. Ελπίζω ότι όσοι ψήφισαν υπέρ της παραμονής θα εξακολουθούν να ε, επηρεάζουν τα πράγματα, αλλά οι άνθρωποι απ' έξω δεν γνωρίζουν τι ε, θα φέρει η επόμενη μέρα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις για σας λοιπόν. Ε, δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να αρχίσει πρώτος ημών των δύο κουν. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Είναι πολύ καλές. Όπως είπατε, κάτι όντως αλλάζει και νομίζω ότι και η αντίληψη ε, και ο τρόπος με τον οποίο η Αφρική ε, στρέφεται, βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει. Ε, επίσης έχουν αλλάξει και πλέον υπάρχουν πολλές ε, αμφιβολίες όσον αφορά την στάση και την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Αφρική. Η Κίνα είναι μεγάλος πρωταγωνιστής παίχτης πλέον. Είναι γεγονός ότι έχει φανεί και στα τελευταία χρόνια ότι και στο κέρας της Αφρικής και στο Σάχελ, ε, εμείς ε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις ε, χώρες. Χώρες οι οποίες είναι εταίροι και τις οποίες προσπαθούμε να κρατήσουμε όρθιες στα πόδια τους και μπορούμε ας πούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα είτε ασφάλειας είτε λοιμού κτλ αλλάζει και ε, ε, ε, αλλάζουν πολλά στοιχεία σε αυτές τις περιοχές, αλλά υπάρχει και ένα σταθερός παράγον που είναι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι και θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας και τα επόμενα χρόνια. Όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει μια εξαιρετική έκθεση του Ιδρύματος Μαχίβαν όσον αφορά τις εξελίξεις ε, στην ε, Αφρική και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς ε, είναι να εστιάσουμε σε αυτές τις προβληματικές ας πούμε περιοχές όπου πρέπει να στηρίξουμε τη διακυβέρνηση, την ασφάλεια, την, τις θέσεις απασχόλησης κτλ. Όσον αφορά την ασφάλεια, την σταθερότητα και τους πόρους που ανέφερε η άλλη σας συνάδελφος. Τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε καλύτερα τα στοιχεία αυτά ε, και αυτό αποτελεί και το κύριο μήνυμα της Φεντερίκα Μογκερίνη, δηλαδή να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε καλύτερα να ε, δράσουμε επί τόπου ε, έτσι ώστε ε, αυτή η δράση μας να έχει αντίκτυπο και σε φαινόμενα όπως είναι η μετανάστευση. Και άλλωστε πώς ε, ε, άλλωστε ένα από τα κύρια στοιχεία τα οποία θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε στη διάρκεια της διάσκεψης είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ε, διευκόλυνση για την Αφρική έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Επίσης με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε καλύτερα να διασυνδέσουμε την ανάπτυξη με την ασφάλεια. Όσον αφορά το μέλλον της Αφρικής ε, σε όρους ε, συμπεριληπτικής κοινωνίας νομίζω ότι υπάρχει ε, ότι είναι κυρίαρχα τα κράτη της Αφρικανικής Υπήρου και αυτά θα πάρουν αποφάσεις αλλά εμείς προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε τέτοιες αρχές και ιδέες για συμπεριληπτική κοινωνία και στην οικονομική διάσταση και στην πολιτική εμπλοκή εμείς προσπαθούμε να έχουμε ακριβώς αυτήν την ίδια στάση. Ε, δύο λόγια ε, για το Brexit που είναι το πιο δύσκολο. Η απάντηση που δίνουμε είναι ότι οτιδήποτε κι αν ε, συμβεί εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες στην Αφρική. Βεβαίως όταν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μαζί μας ε, ε, είμαστε πολύ πιο ισχυροί. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ισχυρός παίκτης και πολιτικός αλλά και όσον αφορά τους αναπτυξιακούς ε, πόρους. Αλλά πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι, και να είναι βέβαιοι και οι εταίροι μας στην Αφρική ότι και μετά το Brexit θα συνεχίσουμε την ίδια αναπτυξιακή προσπάθεια ίσως να ξεκινήσω με τα όσα είπε ο Σαλ όσον αφορά τα γεωστρατηγικά στοιχεία. Υπάρχει η Κίνα όντως, υπάρχει και το ζήτημα του Brexit, υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο και αυτό το έχουν καταλάβει και οι συνομιλητές μας. Υπάρχει και μια αλλαγή ε, παραδείγματος από πλευράς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επομένως, ε, βασιζόμαστε στη σχέση μας στην Αφρική, στις δικές μας πολιτικές αναπτυξιακές αξίες και κατάλαβαν και οι αφρικανικοί εταίροι ότι μετά από την μεταναστευτική κρίση ε, υπάρχει και ένα θέμα συμφέροντος, δηλαδή οτιδήποτε συμβαίνει στην Αφρική δεν αφορά μονάχα την Αφρική. Έχει άμεσο αντίκτυπο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ίσως δίνει μια νέα ε, ε, δυναμική ισορροπία ε, ε, επί σειρά δεκαετιών προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την σχέση ο ένας δίνει, ο άλλος λαμβάνει ε, δωρητού και αποδέκτη. τώρα είναι σαφές ότι υπάρχει και συμφέρον από ευρωπαϊκής πλευράς για παροχή αρρωγής στους εταίρους και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί πιο ισορροπημένες προϋποθέσεις για μια εταιρική σχέση. Και αυτή είναι και η διαφορά ανάμεσα σε εμά και άλλους που εμπλέκονται με την Αφρική. Είναι ότι εμείς βέβαια ε, ε, ε, πάντα σεβόμαστε κάποιες βασικές αρχές. Ας πούμε ότι θα πρέπει να αποκτήσουν ιδιοκτησία των αποφάσεων οι χώρες των εταίρων μας στην Αφρική και εν πάση περιπτώσει εμείς έχουμε κάνει την προσπάθεια να δούμε ε, το, ε, χρονο, το, το, χρονοδιάγραμμα, να δούμε το θεματολόγιο, ε, λαμβάνοντας υπόψη και την θέση της ε, Αφρικής. Δεν είμαστε ε, σαν κάποιους άλλους ε, που έχουν το δικό τους θεματολόγιο και παρεμβαίνουν. Δεύτερο στοιχείο, διάσκεψη κορυφής. Έχετε δίκιο ότι η ίδια η διάσκεψη κορυφής είναι ένα αποκορύφωμα. Πολλά ίδια έχουν αποφασιστεί όταν φτάνουμε στη διάσκεψη κορυφής. Ωστόσο, υπάρχει ε, υπάρχει και το εξή. Ε, Συνήθω στη διασκέψη κορυφή ε, γίνονται μεγάλε δηλώσει προθέσεων. Δηλαδή, συζητούμε και δηλώνουμε το τι προτιθέμεθα να κάνουμε. Επομένω, η προετοιμασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θέλουμε να φτάσουμε σε αυτήν τη διάσκεψη με deliverables, με, πραγματικά παραδοτέα, όχι μονάχα με καλές προθέσεις. Θέλουμε να δείξουμε τι ε, μπορούμε να κάνουμε και τι κάνουμε. Δηλαδή ε, υπάρχουν πράγματα σημαντικά και θέλουν που γίνονται και θέλουμε να το δείξουμε. Και κάποια άλλα στοιχεία, η δημογραφία, το δημογραφικό ζήτημα. Νομίζω πως είναι σαφές ότι η Κίνα δεν θα είχε προχωρήσει, δεν θα είχε πρόοδο ή ανάπτυξη αν δεν είχε ακολουθήσει την πολιτική του ενός παιδιού. Επομένως, η δημογραφική τάση στην Αφρική, όταν βλέπουμε ε, την αύξηση, ε, την τρομερή, ε, είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να εξισορροπήσουμε αυτή την τρομερή δημογραφική αύξηση με ε, την ανάπτυξη. Οπωσδήποτε θα πρέπει να μειωθεί ε, η τάση, να μειωθεί σε σχέση με την προβλεπόμενη δημογραφική ε, τάση. Και επομένως στόχος μας είναι οι γυναίκες. Είναι να δώσουμε δύναμη, empowerment στις νέες γυναίκες και στα κορίτσια. Και αυτό γίνεται μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από την απασχόληση όλες οι μελέτες, όλες οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει με τα Ηνωμένα Έθνη κλπ. Ε, το δείχνουν. Ε, ε, είναι κοινός παρονομαστής η, η, δύναμη που πρέπει να αποκτήσουν οι γυναίκες έτσι ώστε να μειωθεί αυτός ο ρυθμός δημογραφικής ανάπτυξης. Εσείς αναφερθήκατε στις γυναίκες στο Κοινοβούλιο. Βεβαίως εμείς Είμαστε και σε διαρκή επαφή με την πρώην συνάδελφό τη Ιβάνα Κορμέρινγκ, η οποία κάνει τρομερή δουλειά. Εάν θέλουμε ε, να επηρεάσουμε ε, την δημογραφική ανάπτυξη, πρέπει να ε, αναφερθούμε στις γυναίκες και τις γυναίκες βεβαίως στα κοινοβούλια και στην πολιτική. Στο κεφάλαιο διακυβέρνηση καθίσταται σαφές ε, ότι είμαστε πολλοί ε, παρόντες και όσον αφορά ε, την κινητοποίηση δημοσίων επενδύσεων αλλά και όσον αφορά την κινητοποίηση και την μόκλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Αυτό που μας ενδιαφέρει βεβαίως είναι και η σωστή διαχείριση έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα και στην ε, σωστή ανακατανομή. Η Ρουάντα όντως είναι καλό παράδειγμα όπως είπατε αλλά δεν υπάρχουν πολλές Ρουάντες στην Αφρική. Είναι λίγοι οι ηγέτες που γνωρίζουν που θέλουν να πάνε. Είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν μια ομάδα ικανών ε, ε, ε υπουργών που ξέρουν ε, τι θέλουν να κάνουν. Ας πούμε, το Μαλάουι είναι ένα καλό παράδειγμα όπου οι παρεμβάσεις μας είναι πολύ εστιασμένες στην δημιουργία ε, συστήματος κοινωνικής ασφάλειας με ένα θεματολόγιο το οποίο το υποστηρίξαμε από την αρχή και το οποίο τώρα προσπαθούμε να διευρύνουμε με ένα άλλο σκέλος, value change, όπου υπογραμμίζουμε και αυξάνουμε την ε, βιωσιμότητα του ε, συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. σας ζητώ πραγματικά να ε, ε, δείτε τα τελευταία προγράμματα που εγκρίναμε στο Μαλάου, κυρίως στο Κουλιμά, ε, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος σύνδεσης της παραγωγής με την ανακατανομή. Στην Αιθιοπία επίσης κάνουμε σημαντικές προσπάθειες και ένα από τα διδάγματα ε, τα οποία έχουμε συμπεράνει με τον Πρωθυπουργό είναι ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν την ε, προηγούμενη χρονιά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι παρότι η Αιθιοπία δεν έχει ε, φυσικούς πόρους, είχε ανάπτυξη αλλά η κατανομή δεν έγινε σωστά αυτού του πλούτου που παρήχθη. Και σε αυτό το σκέλος βεβαίως θα πρέπει να ε, δώσουμε μεγάλη προσοχή όσον αφορά τις ερωτήσεις, ε, τα ζητήματα τα οποία ανέφερε η Μαρία. Οπωσδήποτε ευθεγραμμίζονται ε, στα όσα προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Βεβαίως η μεταποίηση να γίνεται επί τόπου, βεβαίως να δημιουργήσουμε νέες δεξιότητες έτσι ώστε να αναπτυχθεί η τοπική αγορά αρκεί να δει κανείς ε, ε, ε, τις προσπάθειες που καταβάλει ας πούμε ε, η οργάνωση την οποία να βοηθάει ο Πασκάλ Λαμή ακριβώς προσπαθεί να δημιουργήσει πρωτογενείς, δευτερογενείς ε, αγορές και να τις διασυνδέσει. Δεν νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ανταγωνισμός ε, σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά. Ε, υπάρχουν χώρες όπως η Κένια, ας πούμε, που κάνει παραγωγή ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά πράσινα φασολάκια, ας πούμε, της Κένιας, που τα παράγει η Κένια, ειδικά για τα σούπερ μάρκετ Καρφούρ δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα και έχουν βοηθήσει τις τοπικές αγορές. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα καλού ανταγωνισμού. Προφανώς δεν πρόκειται να πιέσουμε προς την κατεύθυνση της μαζικής βιομηχανοποίησης. Ε, μας, ενδιαφέρει, ε, μας ενδιαφέρουν οι μικρές ε, οι μικρές γεωργικές ε, εκμεταλλεύσεις οι οποίες αναπτύσσονται ε, σε τοπικό επίπεδο και που μπορούν πραγματικά να παραγάγουν θετικό αποτέλεσμα και η έρευνα βεβαίως είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το κοινό κέντρο ερευνών έκανε ε, σχετικές έρευνες ε, για την ε, Αφρική. Ασχολείται με την Αφρική πολύ καιρό και εγώ άλλωστε, γι' αυτό τους παρακολουθώ. Είναι εκπληκτικός ο πλούτος των πληροφοριών που έχουν συλλέξει. 30 χρόνια παρακολουθούν ε, την κατάσταση στην ε, Αφρική ε, και πραγματικά η εικόνα, η απεικόνηση που έχουν έχει μια απίστευτα πυκνή κοκομετρία και πραγματικά απεικονίζει με λεπτομέρεια την πραγματικότητα. Όσον αφορά τον Brexit, ο Κούν νομίζω τα είπε όλα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο και να προσθέσω ευχαριστώ. Thank you very much. Just, um... Ευχαριστώ πολύ. Δύο παραδείγματα που θα ήθελα να αναφέρω και σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις σας. Αυτό που αναφέρατε τη δημιουργία και οικοδόμηση ελπίδας ε, ε και την μη οικοδόμηση τυχόν. Είναι και θέμα του ευρωπαϊκού δρόμου, όπω λέει και η κυρία Μογγερίνη πολύ συχνά. Να σα δώσω μερικά παραδείγματα για το τι ακριβώ ε, αποτελεί αυτό τον ε, ευρωπαϊκό δρόμο και έχουμε και κάποιε εμβληματικέ ε, πρωτοβουλίε που βλέπετε και στην ανακοίνωση για την Σύνοδο Ένα από τα ζητήματα είναι ακριβώ το θέμα τη μετανάστευση. Και νομίζω ότι σε αυτό αναφερόταν όταν έλεγε ότι δεν πρέπει να φτιάξουμε τύχη, ιδίω για τους νέους. Θέλουμε λοιπόν μια ισορροπημένη προσέγγιση και αυτή είναι που ε, διαβουλεύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εταίρους του 2015, αυτό που αποκαλείται Σύνοδος Κορυφής της Βαλέτας. Εκεί θα δείτε τις βασικές αιτίες της νόμιμης μετανάστευσης, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και των εγκληματικών ε, ε, σπηρών, ζητήματα επιστροφ, πολιτικής επιστροφής κτλ. Αυτό είναι το παράδειγμα του ενός ε, δρόμου. Κάτι το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ο ευρωπαϊκός δρόμος λοιπόν για το πώς ε, κινούμαστε στα πιο ε, στα, στα τμήματα της Αφρικής που υπάρχει πιο δύσκολη κατάσταση, ε, ασταθής, Μαλή, Σομαλία για παράδειγμα. Εκεί βλέπετε ότι πολλά από τα προβλήματα συνδέονται και με το γεγονό ότι ο κόσμο δεν έχει πρόσβαση σε αναπτυξιακέ ε, ευκαιρίε και δυνατότητε. Επομένω, για τον ευρωπαϊκό δρόμο που λέμε, χρειαζόμαστε ασφάλεια πάνω απ' όλα. Στο Μαλί έχουμε στρατιωτική στήριξη, αστυνομική στήριξη, αλλά και αναπτυξιακή βοήθεια, σταθεροποίηση και ανθρωπιστική αρρωγή. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτός είναι ο ευρωπαϊκός δρόμος που εμείς θέλουμε ε, να προβάλλουμε όταν ε, πηγαίνουμε σε μια τέτοια σύνοδο κορυφής, όπως αυτή που εξετάζουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για την εξαιρετική σας ε, παρουσίαση και με μεγάλο ενδιαφέρον σας παρακολουθήσαμε γιατί μπήκαμε σε μεγάλο βάθος. Κάποιοι συνάδελφοι έπρεπε να φύγουν γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν παράλληλες συνεδριάσεις, ίσως κάποιο έπρεπε να πάει να ψηφίσει. Αλλά γενικά ήταν πολύ καλή συζήτηση και όπως αναφέρθηκε έχουμε και την, ε, την έκθεση πρωτοβουλία στην οποία θα αποστείλουμε. Θέλετε να πείτε κάτι ακόμα? Ναι, να σας ευχαριστήσω ήθελα μόνο και βεβαίως πάντα είμαστε στη διάθεσή σας να ξαναέρθουμε. Να επαναλάβω μόνο κάτι το οποίο υποκούν. Είναι σημαντικό να κινητοποιήσουμε τα κάτι μέλη μας και νομίζω ότι εσείς έχετε έναν ε, ρολοκλειδί να διαδραματίσετε σε αυτό το επίπεδο, ότι μόνο συλλογικά μπορούμε ε, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με τις σχέσεις μας με την Αφρική. Αυτό γίνεται και με τα Εθνικά Κοινοβούλια, λέει ο Πρόεδρος. Ίσως όταν έχουμε τις επαφές με τα Εθνικά Κοινοβούλια να μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα της Αφρικανικής Στρατηγικής. Συνήθως έχουμε ε, τους ε, προέδρους των αναπτυξιακών επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων αυτοί έρχονται εδώ. Ε, στο Λουξεμβούργο, πρόπερτς, ε, είχαμε κάνει μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων. Ίσως μπορούμε να το σκεφτούμε και αυτό, να προσθέσουμε δηλαδή και την ε, στρατηγική ΑΦΚΟ σε αυτή την συνεδρία. Κάποια στιγμή το φθινόπωρο θα γίνει. Και έτσι να ζωντανέψει και λίγο συζήτηση. Να γίνει λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Για να αξίζει τον κόπο και για εκείνους να έρθουν μέχρι τις Βρυξέλλες. Για εκείνο το έργο στο Μαλάουι μπορείτε να μας στείλετε περισσότερες ε, πληροφορίες. Θέλουμε να ακούσουμε ε, κάτι παραπάνω για τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah, I can say, yeah. So, thank you, colleague. Our next item. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Το επόμενο ζήτημα θα το εξετάσουμε και κλεισμένο των θυρών. Μπορούν λοιπόν να παραμείνουν τα μέλη, οι βοηθοί, συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και γραμματεία. Αλλά δεν είναι δημόσια συνεδρίαση. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αποχωρήσουν.